Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα πρώτα να καλωσορίσω. Uh, dear guests, it is my pleasure to be able to welcome. Ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς και ε, πολλοδεμανό που είστε πολύ άριθμοι. Σας καλωσορίσω στο δεύτερο τμήμα της ε, διακοινοβουλευτικής διάσκεψης ε, με θέμα τους νόμους διάβλους και την ένταξη. Τι γίνεται με όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε, το πρωί είχαμε καταρχήν τη γενική διάσκεψη δύο χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση. Κάναμε ένα απολογισμό της κατάστασης. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για τους νόμους διάβλους και την ένταξη που δεν ήταν ε, ως, δεν ήταν βασική προτεραιότητα της ανταπόκρισης της αντιμετώπισης κρίσης. Ε, μετά μιλήσαμε για το θέμα του, τον νόμο στα πλαίσια του ασύλου και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη διαχείριση της μετανάστευσης και για τους ε, πρόσφυγες και για τους οικονομικούς ε, μετανάστες. Και με αυτή την άποψη η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και με τους πλέον ευάλωτους θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των λύσεων που θα διαλέξουμε. Επίση, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των χρηζόντων προστασία και όσων έρχονται στην Ευρώπη για να εργαστούν. Και αυτό είναι κάτι που το είπαμε με τις Κέγκε στην κοινή μας έκθεση για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε πριν από δύο χρόνια. Και θα προωθήσουμε αυτό το θέμα. Και σίγουρα χρειαζόμαστε και μετανάστες για εργασία. Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, αλλά τα κράτη-μέλη λέμε στην έκθεση ότι θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο τη αγορά εργασία του και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δουν πώ θα γεφυρώσουν τα κενά και θα πληρώσουν τα χάσματα τη αγορά εργασία. Επίση εδώ θα πρέπει να εξάρουμε τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίση, η μετανάστευση λόγω εργασία ε, ε, είναι η διαθέτηση των νόμων διάβλων της νόμιμης μετανάστευσης για οικονομικούς σκοπούς. Επίσης, ε, έχουμε και τα θέματα της ε, διεθνούς προστασίας ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Και ακούσαμε κάποιες ιστορίες φρίκης εκμετάλλευσης ή κακοποίησης των δικαιούχων από την άποψη αυτή και όλα αυτά τα εκμετάλλευση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νομοθεσία στο τομέα αυτό ώστε να ενερμονίσει το νομικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών και το κοινοτικό και εκτιμένο στα θέματα μετανάστευση και λογαγωγού εργασία είναι τομεακό, κλαδικό και δεν υπάρχει ένα ενιαίο κώδικα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλέ και διάφορε οδηγίε που διέπουν διαφορετικά είδη εργαζομένων. Υψηλή ειδίκευση εποχικών, ε, αποσπάσει εντό του ομίλου, ερευνητέ, ε, οπέρ, ε, φοιτητέ. Μόνο νομοθετικό κείμενο που τη χάνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή είναι η αναθεώρηση τη οδηγία για την μπλε κάρτα. Ε, για να προσελκύσουμε ταλέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση, το βασικό μας εργαλείο είναι μία οδηγία του 2003. Στο πάνελ στο οποίο θα προεδρεύσω μέχρι τις 3.30, οι καλεσμένοι μας και τα θέματα που θα πραγματευτούμε είναι αρκετά ευρεία, αλλά κρίσιμα για να προβλέψουμε το μέλλον της ε, διαχείρισης της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα και να δούμε πώς αυτή η διακυβέρνηση, η διαχείριση της ε, ε, μετανάστευση θα συμβάλλει στην οικονομία και τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Κουρτέ είναι διευθύντρια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και θα έχει το δύσκολο έργο να μας παρουσιάσει τις απόψεις ε, της ε, ΠΟΕ της ΔΟΕ μάλλον στο ευρύ θέμα των κενών και των προοπτικών των νομιμών διάβλων στην μετανάστευση για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν ο κ. Τόμας Χάντελσον από το Think Tank, ομάδα μεταναστευτικής πολιτικής, θα μας ενημερώσει για την άσκηση των δικαιωμάτων της οικογενειακής επανένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσαμε και βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα μας παρουσιάσουν την εθνική προοπτική και θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον κύριο Κουζέμπα από την Πολωνική Κάτω Βουλή. Θα ακολουθήσει συζήτηση με συμμετοχή Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών και όπως και το πρωί να κάνουμε κάποιες οργανωτικές ρυθμίσεις. Θα δίνουμε εναλλακτικά το λόγο σε δύο εθνικούς βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή. Θα λαμβάνουν εκ περιτροπής το λόγο μέχρι ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των αγορητών και όπως και το πρωί. Όσοι εθνικοί βουλευτές θέλουν το λόγο του θερμό παρακαλώ να συμπληρώσουν το σχετικό δελτίο, το σχετικό έντυπο και να το χειρίσουν στη γραμματεία που θα τα συγκεντρώνει. Ο κατάλογος των αγορητών θα καταρτιστεί ανάλογα με την σειρά με την οποία έχετε υποβάλει τα αιτήματά σας για αγόρευση. Ενώ οι ευρωβουλευτές μπορούν να μου κάνουν ένα νεύμα ότι θέλουν να μιλήσουν. Και ανάλογα με το χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας και τον αριθμό των επίδοξων αγορητών, θα περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού σε τουλάχιστον δύο λεπτά το χρόνο αγόρευσης και θα σας κάνω νόημα όταν υπερβαίνετε αυτό το όριο. Κυρία Κουρτέγια, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όπως είπατε, η παρουσίασή μου θα εστιαστεί κυρίως ε, στην ε, μετανάστευση για την εργασία και όχι τόσο στους πρόσφυγες. Ο κόσμος πάντα μετανάστευε και θα συνεχίσει να μεταναστεύει. Γιατί ο κόσμος μας είναι όλο και πιο πολύ συνδεδεμένος όσο τα αγαθά και υπηρεσίες ε, διασχίζουν τα σύνορα πιο πολύ παραποτέ, οι ε, τρέχοντες, ε, τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία για του μετανάστε, ο αριθμό δηλαδή των συνολικών μεταναστών, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί. Και αυτό λοιπόν θα χαρακτηρίσει και το μέλλον μα, η μετανάστευση, όπω και το παρελθόν και το παρόν μα. Στην έκθεση των τελευταίων μηνών, ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τόνισε ότι η συνολική μετανάστευση είναι υποφελή και για του μετανάστε αλλά και για τι κοινωνίε που του υποδέχονται. Τόνισε ωστόσο παράλληλα ότι υπάρχουν ε, και λογικά ζητήματα, εύλογα ζητήματα ανησυχία που προκύπτουν από την μετανάστευση, η ασφάλεια, η ξενοφοβία, ρατσισμό, η εντάσει στην κοινωνία. Ε, και για να α, μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στι ανησυχίε αυτέ, ε, ο ΙΕ έχει ζητήσει για να υπάρξουν τακτικέ ε, και ελεγχόμενε μεταναστευτικέ ροέ, οι οποίε θα λάμβανουν χώρα σε ένα πλαίσιο διεθνού δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μετανάστε θα πρέπει να χρησιμοποιούν από πλευρά του τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και να κινούνται τακτικά και οι κυβερνήσεις όμως θα πρέπει και αυτές να ανοίγουν τις οδούς κανονικής και τακτικής μετανάστευσης για να ανταποκριθούν στις πραγματικότητες της αγοράς εργασίας. Γιατί η άτακτη, αν θέλετε, μετανάστευση αυξάνεται όπου υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας και δεν υπάρχει επαρκής ροή μεταναστών αυτή ε, η παράτυπη λοιπόν αυτή η μετανάστευση ε, γεννάται από την ε, ανεπαρκή ροή τακτικών ε, τακτικής μετανάστευσης. Οι ελλείψεις στην αγορά εργασία εντοπίζονται όχι μόνο σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης. Υπάρχουν και πολλές χαμηλή εξειδίκευση ε, δουλειέ, τι οποίε δεν είναι διατεθειμένοι να κάνει το τοπικό εργατικό δυναμικό. Επίση, ε, δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τι τρέχουσε ελλείψει στην αγορά εργασία, αλλά και τι μελλοντικέ που πρόκειται να ανακύψουν σύντομα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία ε, σε ό,τι αφορά τα συμμετέχοντα μέλη που είναι κυβερνήσεις, ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων έχει εκδώσει δύο συνθήκες του 97 και του, και του 143 που έχουν να κάνουν με τις μετανάστες. Ε, φυσικά ε, όλες οι συνθήκες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας σχετίζονται και αφορούν τους μετανάστες. Και πρόσφατα εγκρίθηκε μία σειρά μη δεσμευτικών μέτρων για την πρόσβαση προσπάτως, για παράδειγμα, των μεταναστών και των ε, εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στην αγορά εργασία. Αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2016 από κυβερνήσει, εργαζομένου και εργοδότε και αποτυπώνουν την ε, τριμερή αυτή προσέγγιση για τη μετανάστευση, τονίζοντα το ρόλο που μπορεί να παίξουν οι ε, κοινωνικοί εταίροι στο, στην διαχείριση της μετανάστευσης. Στην καρδιά λοιπόν των συνθήκων και των εργαλείων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας είναι η ίση αντιμετώπιση και η ίση όρια εργασίας μεταξύ των μεταναστών, δηλαδή και του τοπικού πληθυσμού. Αυτή η αρχή είναι κρίσιμη για να εξασφαλιστούν εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και ότι δεν θα υπονομεύονται τα εθνικά πρότυπα ε, εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη οι μετανάστες εργαζόμενοι τείνουν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι η γεωργία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Ο τομέα εστίασης. Αυτή είναι η τομή όπου υπάρχουν και πιο επισφαλείς όροι εργασίας. Άρα, για να είναι ομαλή η μετάβαση και η ένταξη στους τομείς αυτούς, καλό θα ήταν να ενισχυθούν οι θεσμικά όργανα Τη αγορά εργασία, όπω είναι η κατατομή οι ενώσει εργοδοτών, οι εργασία σε οι συλλογικέ συμβάσει κ.ο.κ. Και, και κλείνοντας να πω ότι ανοίγοντα, ε, νομιμέ οδού οδούς δεν είναι μόνο ε, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την ε, κανονική και τυπική σωστή νόμιμη μετανάστευση. Είναι και ένα προαπαιτούμενο προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες ε, επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Και τώρα να βάζω το λόγο στον κύριο Χάτελστον. Για 10 λεπτά κι αυτός. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Λέγομαι Τόμας Χάτελστον από την Ομάδα για τη Μεταναστευτική Πολιτική. Είμαστε ένα think tank το οποίο όμως πράττει κιόλα ε, και δραστηριοποιείται εδώ και πολύ καιρό, κάνει αναλύσεις και αξιολογήσεις για την ε, μετανάστευση και τις ε, διακρίσεις. Με κάλεσαν εδώ για να σας ε, επικαιροποιήσω λίγο τα στοιχεία για την επανένωση των οικογενειών, που είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι ε, μη υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω κάποια σύντομα στατιστικά στοιχεία και μετά κάποιες αλλαγές πολιτικής που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Θα σας πω για τον αντίκτυπο στη μετανάστευση, για την ένταξή τους και τι σημαίνει αυτό για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Καταρχάς, από τότε που ξεκίνησε ο μεγάλος αριθμός των αφήξεων από το 2015, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ε, προσφέρει κάποιο καθεστώς προστασίας σε πάνω από ένα εκατομμύριο υπηκόους τρίτων χωρών. Οι περισσότεροι από αυτούς χρειάστηκαν να έρθουν μόνοι τους, χωρίς την οικογένειά τους, ε, λόγω της έλλειψης ε, ασφαλών διόδων για την έλευσή τους στην Ευρώπη. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να φανταστεί ότι πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Ε, υπήρχαν ε, αφήξεις μεγάλης κλίμακας από το 2015 και τούδε και ε, οι περισσότερες από αυτές ήταν ε, μη προγραμματισμένες, αυθόρμητες, παράτυπες και όχι τόσο ασφαλείς. Η επανένωση των οικογενειών είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Είναι η δυνατότητα οι χώρες ε, να προσφέρουν ασφαλείς, ε, νόμιμες και τακτικές διόδους ε, για τη μετανάστευση. Η επανένωση των οικογενειών ε, γίνεται με αιτήσει, ε, οι οποίε συνήθω ε, διεκπεραιώνονται σε ένα διάστημα έξι μηνών έω ενό έτου. Ε, συνήθως ο μετανάστης έχει ήδη νόμιμη διεύθυνση, γνωρίζει τη σύνθεση της οικογένειάς του και έτσι οι αρχές έχουν αρκετό χρόνο ώστε να φροντίσουν ότι θα υπάρχει κατάλληλη στέγαση και να υποδεχθούν αυτές τις οικογένειες, να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει κατάλληλος χώρος και σχολεία για τα παιδιά και ένα κατάλληλο πρόγραμμα ένταξης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε την επανένωση των οικογενειών με τον ίδιο τρόπο που εξετάζαμε τις ε, αυθόρμητες αφήξει ε, των ανθρώπων που έκαναν αίτηση ασύλου πριν από λίγο καιρό. Ε, δυστυχώς όμως τα τελευταία δύο χρόνια αυτό συνέβαινε. Μέχρι πρόσφατα τα κράτη-μέλη είχαν σχεδόν αντίστοιχε πολιτικές για την επανένωση των οικογενειών και των μεταναστών αλλά και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Για τους μετανάστες ε, ε, διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές έλειπαν πληροφορίες ε, και κάποια στοιχεία ήταν αρκετά περιοριστικά, αλλά για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας τα προβλήματα ήταν περισσότερο ε, τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να διαθέτουν ή ε, τις επαχθές διαδικασίες. Από το 2016 όμως, κάποια κράτη-μέλη ε, είχαν κατηγορηματικές καθυστερήσεις και απεκλεισμό ε, δυνατότητας επανένωσης οικογενειών για άτομα τα οποία την χάνουν διεθνούς προστασίας ή για συνόδευτους ανηλίκους και Μέχρι τότε οι πρόσφυγες, αυτοί οι οποίοι είχαν επικουρικούς προστασίας και ασυνόδευτοι ανήλικοι, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ανα πάσα στιγμή ε, για την επανένωση με την οικογένειά τους. Είχαν καλύτερες συνθήκες από τους ε, υπόλοιπους υπηκόους τρίτων χωρών, είτε για μόνιμες είτε για μακρές περιόδους. Ε, αυτό για την επανένωση των οικογενειών, για του άτομα τα οποία την χάνουν διεθνού προστασία και την περασμένη δεκαετία είχαν μια σταθερή πορεία και μια εύκολη διαδικασία. Από το 2016 όμω και μετά, ε, ένα μεγάλο αριθμό χωρών υποδοχή ε, επέλεξε να επιβάλλει τι λεγόμενε προσωρινέ περιοριστικέ διατάξει, όπου ο λόγο, όπω αναφέρθηκε, ήταν για να μειώσουν ή να καθυστερήσουν τι επανενώσει οικογενείων ε, ή να αποτρέψουν πιθανού περισσότερους ετούντες άσελο. Έτσι είχαμε περιοριστικέ πολιτικέ, οι οποίε είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε πολλέ περιπτώσει δεν τι είχαμε ξαναδιαπιστώσει. Αυτοί οι περιορισμοί ε, ε, επιβλήθηκαν στην Αυστρία, στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στη Δανία και στη Σουηδία. Οι περιορισμοί λοιπόν ε, επρόκειτο να είναι προσωρινά μέτρα, αλλά πολλοί από αυτού εξακολουθούν να ισχύουν, παρά το γεγονό ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τελείω διαφορετική κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για εσά, ω πολιτικοί ηθήνοντε, να αντιληφθείτε ότι η επανένωση των οικογενειών θα πρέπει να την χάνει διευκόλυνση σε όλα τα κράτη-μέλη ε, καταρχάς, ε, διότι όταν εξετάζουμε την ένδειξη των μελών τη οικογένεια, ε, βλέπουμε ότι η διαδικασία είναι μεν χρονοβόρα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία τη Eurostat αποδεικνύουν ότι μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια στη χώρα, η πλειοψηφία των μελών ε, μια οικογένεια που έχουν συναντήσει τον πρώτο υπήκο, έχουν ενταχθεί και έχουν θέσει εργασία. Προσφέρεται δηλαδή χρόνο και στήριξη για την επανόνωση των μελών τη οικογένεια. Πολλέ, για παράδειγμα, σύζυγοι ορισμένες φορές έχουν απλώς ε, πολύ γενικά προγράμματα ένταξης που δεν είναι τόσο αποτελεσματικά για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι χώρες δεν έχουν βελτιώσει και τόσο πολύ τις πολιτικές ένταξης και τα προγράμματά τους ε, για τις συζύγους αυτές. Επιπλέον, η στήριξη που προσφέρεται για τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα επίσης δεν έχει βελτιωθεί ε, σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αργούν συνήθως να εφαρμόσουν ε, τα μέτρα στήριξης που χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό οι πολιτικές ένταξεις και οι διαδικασίες να βελτιωθούν τόσο για τις ε, συζύγους αλλά και για τα παιδιά τους. Ε, δεν είναι όμως το μόνο στοιχείο στο οποίο επικεντρωθήκαμε. Ε, όπως διαπίστωσα, πολλές από τις αλλαγές της πολιτικής ήταν περισσότερο περιορισμοί ή καθυστερήσεις στη διαδικασία της επανένωσης και η έρευνα καταδεικνύει ότι αυτές οι καθυστερήσεις ουσιαστικά βοηθούν να καθυστερήσουμε και να υποσκάψουμε την όλη διαδικασία ένταξης και για τον ε, χορηγό, ο οποίος ε, μπορεί και να ε, πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας ακριβώς λόγω της καθυστερήση, αλλά και για τους τις συζύγους και τα παιδιά. Διότι αυτοί οι περιορισμοί απλώς ε, ε, καθυστερούν τη διαδικασία ένταξης. Για παράδειγμα, η μελέτη της πίζας του ΟΣΑ ε, διαπίστωσε ότι κάθε χρόνο επιπλέον που τα παιδιά πρέπει να περάσουν στη χώρα καταγωγής τους ε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μάθουν τη γλώσσα και θα αριστεύσουν στο σχολείο στη νέα χώρα. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Όσο περισσότερο υποχρεώνονται οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στις χώρες καταγωγής τους, τόσο λιγότερο χρόνο έχουν για να έρθουν σε επαφή με τα δικά μας τα όργανα και τα δικά μας εκπαιδευτικά συστήματα. Τα παιδιά δηλαδή φτάνουν στη χώρα σε μεγαλύτερη ηλικία και δυσκολεύονται να ενταχθούν περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για συζύγους που δεν είναι σε θέση ε, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ε, και ε, φυσικά να μάθουν και γλώσσα όπως και ο πρώτος Ε, και βλέπουμε λοιπόν ότι δυσχεραίνονται τα αποτελέσματα της ένταξης ακριβώς λόγω των καθυστερήσεων αυτών. Αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος διέπεται ούτως ή άλλως ήδη από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υπάρχει η Οδηγία Επανένωση των Οικογενειών του 2003-86 και είναι και ένας τομέας ο οποίος ρυθμίζεται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Ε, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει διευκρινίσει ότι η οδηγία για την επανένωση των οικογενειών έχει ως πρωταρχικό στόχο να διευκολύνει την οικογενειακή ζωή και να προωθήσει την επανένωση της οικογένειας. Βάσει αυτής της νομολογίας, οποιαδήποτε διάταξη επανένωσης οικογενειών πρέπει να είναι ε, δεόντως αιτιολογημένη, αναλογική και αποτελεσματική. Θεωρώ λοιπόν ότι ήγηκε η ώρα να ε, επανεξετάσουμε τις περιορισμούς αυτούς για την επανένωση των οικογενειών που εφαρμόστηκαν ίσως ε, κάποια στιγμή που ε, είχε επικρατήσει ο φόβος και το άγχος και πλέον θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτές τις πολιτικές για να διευκολύνουμε την ταχεία επανένωση των οικογενειών για συζύγους και παιδιά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Και για να τονίσουμε πλέον τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο αποτελεσματικά προγράμματα ένταξης ε, για συζύγους και παιδιά. Ε, αν θέλετε κάποια περισσότερα για τα θέματα αυτά, θα ήθελα να σας συστήσω να δείτε τον δίκτυ πολιτικής ε, ένταξης ε, της μετανάστευσης. Επίσης να δείτε την πρόβλεψη του 2017 του ΟΣΑ για τη διεθνή μετανάστευση που έχει όλα τα στοιχεία για τις πιο πρόσφατες αλλαγές πολιτικής. Επίσης να διαβάσετε τις συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης του 2017 το οποίο αφορά συγκεκριμένα την επανένωση οικογενειών και επίσης συστήνω να εξετάσετε ή να μιλήσετε με το, τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Νίλ Νιούσνικ, ο οποίος έχει δημοσιεύσει πολύ ε, καλά έγγραφα, δύο πολύ καλά έγγραφα, πολύ ευανάγνωστα, ε, που μπορείτε να τα δείτε και τι, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει για την επανένωση οικογενειών για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάτσομ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κουζέμπα από την Πολωνική Βουλή που θα μας παρουσιάσει την ε, εθνική προοπτική και την κατάσταση στην πατρίδα του, την Πολωνία. Σας ευχαριστώ, σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω μάλλον ε, εγκάρδια. Ε, πολύ εντυπωσιακή η συζήτηση και θα ήθελα να σας παρουσιάσω και κάποια πολωνική θεώρηση και το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στη δική μας χώρα. Πολύ συχνά επικρατεί μια τοπική θεώρηση και αυτό μας δημιουργεί μια περιορισμένη προοπτική και αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την ευεργεσία που προσφέρουν άλλες χώρες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις, τη δυνατότητα που μας δώσετε να ακούσουμε αυτές τις ομιλίες ε, και από τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Ουγγαρία ε, και θα αναφερθώ και σε μερικά από αυτά που συζητήθηκαν το πρωί. Επίσης, ε, τα έθνη και τα κράτη έχουν τις δικές τους ένομες τάξεις, έχουν το δικό τους νομικό σύστημα, έχουν την ε, εθνική κυριαρχία να διαμορφώνουν το πεπρωμένο τους και αναλαμβάνουν επίσης τις ευθύνες για τα έργα τους, αφήνοντας τη δική τους παρακαταθήκη και δεν θα πρέπει να σφετεριζόμαστε αυτή, αυτά τα προνόμια. Θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερα τα κράτη-μέλη να ασκήσουν αυτή την εθνική τους πολιτική. Επίσης, η πεμπτουσία της ομιλίας μου θα είναι μια παράκληση να σκεφτούμε όλοι μαζί ότι Μερικές φορές είναι εύκολο να εξάγουμε τη βοήθεια, την ευημερία και να στηρίξουμε τα περιβάλλοντα, τις χώρες, τα έθνη στα οποία υπάρχει μια έλλειψη οργάνωσης και ένα χάος. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε εξαγωγή καλού από ότι εισαγωγή ε, προβλημάτων και ταραχών που θα οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερα προβλήματα στο εσωτερικό των δικών μας χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω καταρχήν την παρούσα κατάσταση στην Πολωνία που έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, έχει μια ιδιαιτερότητα. Τα τελευταία χρόνια ε, η Πολωνία μετατράπηκε από ε, χώρα αποδημίας σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ευημερίας ε, και της ένταξής μας το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τότε πολλοί Πολωνοί έφυγαν από την Πολωνία, αναζητώντας ε, αλλού ε, θέση, απασχόληση. Σα απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε για την θερμή υποδοχή που τη επιφυλάξατε, αλλά σκεφτείτε όμως με τι επαγγελματισμό και με τι πολιτιστικό υπόβαθρο ε, βρίσκονται αυτοί οι Πολωνοί στις δικές σας χώρες. Βέβαια, είναι ο μεγαλύτερος απόδημος πληθυσμός της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης είναι ταυτόχρονα και ε, πόλος ε, μετανάστευσης από τις ανατολικότερες της ε, χώρες. Για παράδειγμα, έχουμε μετανάστες από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την Ρωσία, τη Γεωργία, την Αρμενία. Τότε είμαστε πόλος μετανάστευσης και όχι χώρα αποδημίας. Έχουμε λοιπόν απλουστευμένες διαδικασίες για τους μετανάστες αυτών των χωρών για να τους διευκολύνουμε με προσωρινές διατάξεις έξι μηνών. Αυτό έχει και για τη Μολδαβία και στη συνέχεια γίνεται η καταγραφή τους προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν και θέσεις ε, απασχόλησης. Δεν πρόκειται να σας ε, κουράσω με στατιστικά στοιχεία, αλλά ε, λένε πολλά. Το 2016 η Πολωνία για τέταρτη συνεχή χώρα, χρονιά είναι η δεύτερη χώρα μετά τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αδειών, δηλαδή 580.000 περίπου άδειες Επίσης, ε, για τις μακροχρόνιες ε, επισκέψεις, 17% όλων των αδειών παραμονής ε, που εκδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις άδειες εργασίας, η Πολωνία βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις θέσεων αδειών εργασίας. 494.000, δηλαδή σχεδόν μισές από αυτές που εκδίδονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η στην Πολωνία έχουμε περισσότερο, ε, περισσότερους Ουκρανούς. 17,5% των ε, αδειών ε, ολόκληρης Ευρώπης βρίσκονται στην Πολωνία. Και 81% ε, από αυτές τις 500.000 άδειες εκδίδονται στην Πολωνία. Επίσης, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία Ουκρανών μεταναστών στην Πολωνία. Ε, ο αριθμός των μεταναστών που απασχολείται στην Πολωνία αυξάνεται συνεχώς. Και μάλιστα η στριπτική της ψηφία ε, ε, ακολουθούν απλουστευμένες διαδικασίες και μπορούν για τρεις μήνες να εργάζονται χωρίς άδεια και μετά για 12 μήνες μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους αρκεί να είναι εγγεγραμμένο το γραφείο στο οποίο απασχολούνται. Σας δίνω όλα αυτά τα στοιχεία με την ελπίδα ότι θα εκτιμήσετε το μόχθο της Πολωνίας και τις προσπάθειες που καλείται να κάνει αυτή η χώρα με αρκετή ε, διαλλακτικότητα, με μεγάλο άνοιγμα προς τους χιλιάδες ε, μετανάστες της Ανατολικής Ευρώπης, του πρώην Σοβιτικού Μπλοκ, που αναζητούν μία θέση εργασίας στην Πολωνία. Τώρα, ως προς την σημερινή συζήτηση, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ευρύτερε προοπτικές. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό πρόβλημα θα πρέπει να εξεταστεί και διαδικαστικά. Θα πρέπει να εξετάσουμε τους παράγοντες και τους μηχανισμούς ε, που διέπουν την παράτυπη και να τη διακρίνουμε από την νόμιμη μετανάστευση των φοιτητών, ερευνητών, εργαζομένων και εποχιακών εργαζομένων. Επίσης υπάρχουν μεγάλες μεταναστευτικές διακυμάνσεις στις μεταναστευτικές ουραίες και μερικές φορές είναι και απρόβλεπτες. Γι' αυτό καλό θα ήταν συνειδητά να καθοδηγήσουμε την νόμιμη μετανάστευση ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και όταν μιλούμε για την ε, μπλε κάρτα θα πρέπει να γίνει μια διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Και από αυτή την άποψη έχουμε τρία πολύ, τέσσερα, ή τρία, τέσσερα πολύ σημαντικά θέματα και ζητήματα. Γιατί η διάγνωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί. Και η συγκεκριμένη διάγνωση της αγοράς εργασίας θα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα, ανάλογα με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Και από αυτή την, άπτωση, από αυτή την άποψη έχουμε διαφορές ε, ε, σε ό,τι αφορά και τους εργοδότες και τις ανάγκες των εργοδοτών. Θα πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ των χωρών που, έχουν, ε, τους, που εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους και για πολύ φυσιολογικούς και εύλογους τρόπους. Αυτός ο εργαζόμενος που έχει εκπαιδευτεί, που έχει σπουδάσει σε μια χώρα, αποδημεί σε άλλη χώρα για να βρει καλύτερη θέση απασχόλησης. Για παράδειγμα η Πολωνία, η Τσεχία, η Γαλλία που επένδυσαν στην εκπαίδευση αυτού του εργαζόμενου. Γιατί να χάνουν τις ειδικότητές του και τις δεξιότητές του όταν αυτός αποδημεί σε άλλη χώρα για να βρει θέση απασχόλησης. Πώς θα αντισταθμίσουν τις επενδύσεις που έκαναν στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση αυτού του εργαζομένου οι χώρες αυτές. Επίσης, ε, έχουμε μία αύξηση ε, τεράστια και της οικονομικής μετανάστευσης και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ε, εργαζόμενους που ήδη έχουν μια θέση απασχόληση δηλαδή και εκείνους που έρχονται με σκοπό να αναζητήσουν θέση ε, απασχόλησης και πώς θα τους ετοιμάσουμε για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Και στο πακέτο αυτό των ζητημάτων, στη δέσμη αυτών των ζητημάτων έχουμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η νέα γενιά των Ευρωπαίων. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της γύρας του πληθυσμού. Είναι πολύ ε, σημαντικό, ένα θέμα που ανακύπτει, το θέμα της κατάστασης της αγοράς εργασίας και το πρόβλημα της ε, δημογραφικής παρακμής ε, λόγω της γύρας του πληθυσμού. Ενώ ταυτόχρονα σε μερικές χώρες έχουμε υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων. Οπότε θα είναι λογικό να ανακύψει το ζήτημα πώς ε, θα αξιοποιήσουμε σωστά τις νέες γενιές και θα τους ε, δώσουμε ένα ευρύ φάσμα ε, επαγγελματικής ε, διεξόδου και σταδιοδρομίας. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των εργαζομένων που στην Πολωνία, που σήμερα είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία, οι εργαζόμενοι στην Πολωνία ίσως έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ε, επαγγελματικά από ότι ε, οι εργαζόμενοι που αναμένονται στην Ολλανδία. Και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή έχουμε ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών μελών για την προσέλκυση εργαζομένων. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη διαδικασία επιλογής των εργαζομένων για τις αγορές εργασία. μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κουζέμπα. Θα περάσουμε στη συζήτηση με τους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο-τρία λεπτά ο καθένας. Και επίσης να υπενθυμίσω στους βουλευτές που θέλουν το λόγο να μην ξεχάσουν να συμπληρώσουν το έντυπο. Οι κλητήρες κυκλοφορούν και συγκεντρώνουν τα έντυπα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Φρανκ Τιρτσεκ που είναι Σλοβαίνος βουλευτής. Παρακαλώ. Δεν ξέρω που κάθεστε όμως. άλλαξε ο πρώτος ομιλητής, τότε πείτε μας ποιος είστε. Ναι, σας ευχαριστώ και θα μιλήσω Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι σύντομος στην παρέμβασή μου. να παρουσιάσω λοιπόν τα επιχειρήματα από πλευρά μα. Στη Σλοβενία, η κυβέρνηση. Είναι αριστερή κυβέρνηση. Εγώ είμαι από την αντιπολίτευση, το κόμμα τη αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά δε την στάση της Σλοβενίας εναντί της μετανάστευσης, να σας παρουσιάσω μια πληροφορία η οποία θεωρώ ότι είναι σχετική το 97 Δεχτήκαμε 4% των ε, μάλλον μεταναστών σε σχέση με τον ε, πληθυσμό τη Σλοβενία, 4% μετανάστε. δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Ήταν κυρίω γυναίκε, ε, ε, πιο ηλικιωμένε γυναίκε, παιδιά, ηλικιωμένα ως επιτοπλίστων άτομα, τα οποία ήλθαν στη Σλοβενία μέσω την οδού των Βαλκανίων και το 2014-2015 οι μετανάστες ήταν κυρίως νεαροί άντρε, Δεν είναι πλέον γυναικόπαιδα. Η σλοβανική κυβέρνηση λοιπόν συμμετέχει στο σύστημα των ποσοστώσεων όπως αποκαλείται και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υποδεχόμαστε και μετανάστες από την Ελλάδα και την Ιταλία. Τα νούμερα είναι χαμηλά σχετικά γιατί είναι μικρή η χώρα μας. Ωστόσο, πέρσι σημειώθηκε αύξηση 1300%, 1300 σε ό,τι αφορά την υποδοχή μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας εγκομιάζει και ο Πρωθυπουργός έχει υποφεληθεί σε διάφορες φωτογραφίσεις και φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και λειτουργούν σωστά. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αυτών, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που κατέφτασαν στη Σλοβενία, είτε ήταν τμήμα των μεταναστευτικών ροών, είτε απεστάλησαν στην Σλοβενία στο σύστημα των ποσοστώσεων. 80% των ανθρώπων αυτών ήταν στη Σλοβενία ως χώρα Διέλευση. Έφυγαν δηλαδή και από τη Σλοβενία μέσα σε λίγε μέρε. Το σύστημα των ποσοστώσεων λοιπόν φαίνεται ότι λειτουργεί. Δεν λειτουργεί όμω στην πράξη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τι χώρε μόλι καταχωριστούν στο σύστημα. Άρα το σύστημα δεν θεωρώ ότι λειτουργεί όπω θα έπρεπε. Θα πρέπει να βρούμε καλύτερε λύσει πιο σωστέ και αποτελεσματικέ. Εγώ προσωπικά έχω ορισμένε υπόψη μου. Καταρχάς, όπως είπαν και συνάδελφοι από την Τσεχική Δημοκρατία, από τη Σλοβακία, από την Ουγγαρία. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις χώρες εκείνες όπου επικρατούν συγκρούσεις οι οποίες και προκαλούν τη μετανάστευση. Αυτό ασφαλώς αποτελεί σημαντικό στόχο. Περαιτέρω όμως θα πρέπει να επιτηρούμε και να προστατεύουμε τα σύνορά μας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν συμφωνώ με όσους θέλουν να αλλάξουν οι κανόνες. Να αλλάξουν οι κανόνες για να μετατραπεί η παράνομη μετανάστευση σε νόμιμη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε καλύτερε λύσει, θεωρώ, που θα ωφελήσουν, θα ωφελήσουν πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς. Και την ίδια την Ευρώπη. Ανέφερα ήδη κάποιε από τι λύσει αυτέ. Δεν έχω ωστόσο χρόνο για να περάσω σε μεγαλύτερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μέτσολα. Ήσασταν, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τούτσεκ αργότερα. Η επόμενη ή ο επόμενο. Ο κύριο Ζάκλιν από την Γερμανική Βουλή. Από το Γερμανικό Bundestag. Η κυρία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Νάστεκ. Είναι θετικό το γεγονό ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά κανενό ε, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και ότι θα πρέπει να τηρούνται οι ίδιοι εργασιακοί όροι. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από Πρακτική πλευρά και από πολιτική πλευρά, Είτε πρόκειται για εργοστάσια μεταποίηση ε, ε είτε πρόκειται για τον τομέα τη νοσηλείας. Και επίση ε, υπάρχει η κατάχρηση των μεταναστών από τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις, από του μεγάλου ομίλους. Αυτό δημιουργεί ασφαλώ και κακή ε, ατμόσφαιρα κατά των μεταναστών. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία και η ξενοφοβία κατά των ε, Πολωνών που αυξάνεται. Στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, είπατε. Εγώ διαφωνώ. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, την οδηγία για την μπλε κάρτα, θα πρέπει να φροντίσουμε σε ό,τι αφορά να μην καταλήξουμε σε dumping μισθών, να μην καταλήξουμε σε μείωση των εργασιακών συνθήκων Μήπως ε, ε, αυτό τελικά θα καταλήξει να οδηγήσει σε μια κατάσταση των ε, εταιριών, σε brain drain, διαρροή και διαφυγή των επιχειρήσεων και των εγκεφάλων. Θα πρέπει στόχος να είναι η ενισχύση της τοπικής μηχανίας, η υποστήριξη ιδιαίτερως των φτωχών χωρών. Ρωτώ λοιπόν με ποια μορφή θέλετε να υποστηρίξετε την εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό στις χώρες προέλευσης για να μην γίνουν ακόμα πιο φτωχές αυτές οι χώρες και να μην γίνεται μόνο επιλογή προς όφελος του κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις οικογένειες, να πω δύο λόγια, συζητιέται στην παρούσα φάση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο το θέμα της, της ε, οικογενειακής επανένωσης και αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ενσωμάτωσης και ασφαλώς είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε. Δυστυχώς όμως ε, ο συνασπισμός των κυβερνών στην ε, Γερμανία τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εμείς ως αριστερά θέλουμε να υπάρχει καλή ενσωμάτωση, ιδιαίτερα για την ετήρηση της αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I Σας ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από το ΕΛΚ, τον κύριο Μπονή. Θα μιλήσω πολωνικά. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την διοργάνωση της σημερινής διακοινοβουλευτικής διάσκεψης και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Γιάτσε Κουζέμπα, ο Πολωνός βουλευτής. Ήταν πολύ λογικά όλα αυτά που μας είπε, πολύ συνετά και πολύ σωστά προσέγγισε το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης. Βέβαια, στην Πολωνία έχουμε και μία μεγάλη ομάδα Ουκρανών κυρίως πολιτών που νόμιμα απασχολούνται στην ε, Πολωνία και πέρυσι το 2017 εκφράστηκε η ανησυχία όταν ε, απελευθερώθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίου για τους Ουκρανούς για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε κάποιος φόβος, αλλά ήδη έχουν περάσει εννέα μήνες και δεν είναι ότι αφήνουν τις θέσεις εργασίας τους στην Πολωνία και τρέχουν προς την Γερμανία να απασχοληθούν οι Ουκρανοί όπως αρχικά είχε ε, διαρρεύσει ένας φόβος. Και σίγουρα η σχέση με τις γειτονικέ χώρες στο, πλαίσιο, στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης είναι πολύ σημαντική. Και σίγουρα ε, ε, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, κάθε χώρα έχει απλουστευμένες διαδικασίες. Ίσως για μερικούς τομείς ε, θα μπορούσαμε να απλουστεύσουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες και όταν ε, ξεκινούμε κάποιες διαδικασίες ένταξης, είναι σημαντικό να τις λάβουμε αυτές τις διαδικασίες ένταξης ευρύτερα, καλύπτοντας και τα παιδιά, ώστε να μπορούν να φοιτούν στα σχολεία και να μην χάσουν την φοιτησή στα πολωνικά σχολεία. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολωνοουκρανικές σχέσεις, ε, η κατάσταση είναι πολύ καλή. Ε, τα παιδιά από την Ουκρανία νιώθουν πολύ καλά στα πολωνικά σχολεία και έχω πολλές μαρτυρίες από φίλους και συγγενείς. Και μάλιστα η Πολωνία είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα της διαμόρφωσης μιας νέας ανοιχτής μεταναστευτικής πολιτικής. Και όπως είπε ο κ. Κουζέμπα, μιλάμε πολύ καθαρά α, για τους μετανάστες και τη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ μετανάστευσης και προσφυγιάς, μεταναστών και προσφύγων. Αυτό το θέμα στην Πολωνία είναι αρκετά επίμαχο και αφιλεγόμενο. Η προσωπική μου γνώση είναι ότι ε, σε πολλές χώρες οι πρόσφυγες γίνονται νόμιμοι μετανάστες, ε, ε, εντάσσονται στην αγορά εργασίας και την εμπλουτίζουν με τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Πάντω αυτό είναι θέμα προσυζήτηση. Σίγουρα η Πολωνία είναι ένα καλό παράδειγμα μεταναστευτική πολιτική και μάλιστα μεγάλη κλίμακο, γιατί μιλούμε για εκατοντάδε. χιλιάδες ε, εργαζόμενου μετανάστε. Επίσης, ε, ο κύριος Κουζέμπα μίλησε για το διαδικαστικό ζήτημα, πολύ σωστό, με ανάμειξη και ευλοκή όλων των ε, κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Ευχαριστώ, Μιχαήλ. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Τσίρτσακ από τη Σλοβενία. Okay, thank you, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στα σλοβενικά. Αρχικά σκόπευα να σας παρουσιάσω την άποψή μου στο επόμενο πάνελ, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να τα πω και τώρα. Δεν είμαι πολιτικός ε, σταδιοδρομίας, ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια την ενασχόλησή μου με την πολιτική και παρακολουθώ στενά το θέμα της μετανάστευσης. Αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα, συζητήσαμε και στα προηγούμενα πάνελ, περιστρέφονται γύρω από το θέμα της πολιτικής οικονομίας. Πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, πρόκειται για οικονομικό ζήτημα στην ουσία του. Εάν ε, εξετάσουμε το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο διαθέτει η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία για την ένταξη των μεταναστών, ε, είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Σε κάποιες χώρες ε, δίνονται πολύ περισσότερα για την ένταξη από ό,τι σε άλλες, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία. Θα επενδύσουμε λοιπόν ε, ε, κάποιες ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερα για να επιλύσουμε το ζήτημα, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό βεβαίως ε, σημαίνει ότι οι μετανάστες θα πρέπει να απολαμβάνουν και τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τη δυνατότητα εργασίας και ε, φυσικά αρκετοί οικονομικοί τομείς επηρεάζονται και από την εμπορία ανθρώπων. Η γεωργία, ο τομέας της στέγασης, ο κατασκευαστικός τομέας ε, και πολλοί άλλοι. Εμείς όλοι είμαστε συνταγματικές δημοκρατίες, αλλά στους τομείς αυτούς ε, το Σύνταγμα παραβιάζεται. Και μάλιστα το θέμα αυτό είναι στο επίκεντρο του προβλήματος. Οι λαϊκιστές κατά πάσα πιθανότητα θα πούνε ότι στη Σλοβενία, στην Πολωνία ή όπου αλλού υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, φταίνουν οι μετανάστες γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Πώς γίνεται κάποιος ε, παράτυπος μετανάστης. Ε, δεν υπάρχει ε, παράνομο άτομο. Μπορεί κάποιος να βρεθεί στην παρανομία όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη χαμηλοι μισθοι φταινει μεταναστες γι η πολιτική είναι διεφθαρμένη και πρέπει να βρεθει στην παρανομια οταν δεν υπαρχει ειλικρινείς μεταξύ μας γιατί όλοι πολιτικοί είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάιερ από τη Γερμανία στη συνέχεια. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. καταρχά σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση, διαπιστώνουμε κυρίω στη Γερμανία ότι έχουμε περίπου 540.000 άτομα τα οποία σύμφωνα με τις συνθήκες της Γενέβης ε, αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες χωρίς να έχουν πλήρες όμως δικαίωμα για οικονομική επινένωση και φυσικά αυτές τις υποχρεώσεις, τις, ε, αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να τα απολαμβάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα περιορισμό. Και μιλάμε λοιπόν για τα άτομα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν τα δικαιώματα αυτά μέχρι 16 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ε, η Γερμανία έχει περίπου 270.000 άτομα τα οποία επικουρικά θα πρέπει να βοηθηθούν, δηλαδή είναι πρόσφυγες ε, και που έχουν σαφείς προσδοκίες σε ό,τι αφορά την ε, υποδοχή τους και τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, θα πρέπει να γυρίσουν επίσης στις χώρες τους μετά τη λήξη των εμφύλιων συγκρούσεων. Εδώ λοιπόν η ενσωμάτωση δεν είναι το βασικό μέλημα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι εγώ και η πολιτική μου, το πολιτικό μου κόμμα, ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε, να σταματήσουμε να κόψουμε την ισχύ των μέτρων αυτών ενσωμάτωσης για τα άτομα τα οποία θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία θα αφορά ε, κατά ελάχιστη κατά το όριο για 12.000 άτομα και θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αντικειμενική και πολύ ανθρωπιστική τέτοια ρύθμιση γιατί έχει να κάνει και με άτομα τα οποία έχουν ε, σημαντικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση τώρα, έχω την εντύπωση ότι συνδυαρκώς κάνουμε το λάθος ε, ότι έχουμε αυτή τη διάκριση, την ανθρωπιστική μετανάστευση, όπου δεν υπάρχει νόρη, και έχουμε και το δεύτερο είδος μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εργατική, εργασιακή μετανάστευση. Η ΕΠΑ ΕΕ είναι η δεύτερη, χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα ε, με την ε, τέτοια εργασιακή νόμιμη μετανάστευση. Δεν μπορεί να είναι όμως ε, σαφές αυτό. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει για να μην είναι πολύ μεγάλη η ενιαία διαμορφώση των κανόνων και τελικά καταλήξουμε να κάνουμε διακρίσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούμε να έχουμε 28 διαφορετικές αγορέ εργασία. και οι ανάγκες είναι διαφορετικές σε κάθε μία εξ αυτών. Και αυτό λοιπόν ζητώ την κατανόησή σας καταπηγόντως ω εθνικοί βουλευτή, θα επιμείνουμε στη θέση μας ότι η εθνική αρμοδιότητα θα πρέπει να μην επηρεάζεται καθόλου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εθνική αγορά εργασία. Η Γερμανία στην παρούσα φάση έχει μια οικονομία η οποία πάει καλά. Έχουμε πλήρη απασχόληση σε πολλά τμήματα τη χώρα και ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ ετερογενή, επαναλαμβάνω, η αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μία ρύθμιση να ισχύει εφάπαξ για 28 διαφορετικές αγορές εργασίας και 28 διαφορετικές οικονομίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πάλης από την Ελλάδα. Καλησπέρα και πάλι. Θα μιλήσω μόνο για το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης. Και θα είμαι σύντομος. Ε, οφείλω να σας πω ότι η στέρηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στους ανθρώπους αυτούς, έναν διπλό εγκλωβισμό. Καταρχήν στα hotspot και στη συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα εισόδου των προσφύγων αυτών. Μιλάμε ουσιαστικά για ανθρώπους που η ζωή τους μπαίνει στο ψυγείο. Και μπαίνει στο ψυγείο για προσδιορίστο χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν έχουν καμία διάθεση εκμάθηση της γλώσσας στη χώρα στην οποία ζουν, εκπαίδευση και ένταξη. Το μόνο που επιθυμούν είναι η γρήγορη οικογενειακή επανένωση. Οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία τραγικές. Έχουν αδυναμία αντίληψη του αυτονόητου, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν με τους δικούς τους, που πολλές φορές τους οδηγεί σε εντός εισαγωγικών εναλλακτικές δράσεις για την διεκδίκηση του, του αυτονόητου δικαιώματος. Μιλάμε δηλαδή για απεργίε πείνα. Είχαμε πρόσφατα το Δεκέμβριο στο κέντρο της Αθήνας απεργία Πείνα προσφύγων που περιμένουν την οικογενειακή επανένωση. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι και απόλυτα κατανοητό νομίζω από όλους μας είναι ότι γι' αυτό το πρόβλημα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό που του συμβαίνει. Δεν φταίει η χώρα υποδοχής, φταίνε οι χώρες που αντιδρούν στην οικογενειακή επανένωση. Εγώ κατανοώντας τον Γερμανό συνάδελφο, Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει το πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι χώρε εισόδου και οι χώρε όπου συντελείται η οικογενειακή επανένωση. Παρόλα αυτά όμω, για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν είναι ο μεγάλο αριθμό, είναι μάλλον ένα μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των προσφύγων, μπορούμε και καλύτερα να δράσουμε και γρηγορότερα με δεδομένο ότι οι συνέπειε τι όλε τι καθυστερήσει μπορεί να είναι χειρότερε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι το ίδιο το αποτέλεσμα τη γρήγορη επανένωση των οικογενειών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μάρεκ Γιούρεκ, σας ευχαριστώ. Przepraszam. prowadzimy Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή και ο διάλογος που έχουμε με τους εθνικούς βουλευτές. Ε, μας δίνουν μια εθνική διάσταση στη συζήτηση, πολύ χρήσιμη. Σε ό,τι αφορά το θέμα της οικογενειακής επανένωσης, θα ήθελα να σταθώ σε ένα βασικό σημείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με μεγάλες παρεμβολές στο μικρόφωνο, δυστυχώς, στο μιλητή. Πριν από 50 χρόνια, η μετανάστευση στη Γαλλία ήταν κυρίως μετανάστευση από τη Νότια Ευρώπη τη δεκαετία του 20, τη δεκαετία του 30, ε, ήταν μετανάστευση από την Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Σήμερα οι μετανάστες στη Γαλλία είναι κυρίως από την Βόρεια Αφρική και την Αιγής Ανατολή, ή τη Μέση Ανατολή. Από το Μαρόκο μέχρι την Ιδονησία έχουμε μια σειρά χωρών που έχουν πολύ διαφορετικά αστικά και οικογενειακά δίκαια και διαφορετικά έθιμα. Για παράδειγμα, έχουν την πρακτική της πολυγαμίας, οπότε από αυτή την άποψη η οικογενειακή επανένωση λαμβάνει διαφορετική χρειά. Επίσης, το θέμα της ύπαρξης ε, των παιδιών. Δεν έχουμε παράνομους ανθρώπους σίγουρα, αλλά ο έλεγχος των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι νόμιμο και αν ε, θεωρεί κανείς παράνομη παράνομο τον έλεγχο των εξωτερικών σύνορων, τότε ε, τι να πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες που εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση ε, στην επικράτειά τους και κάποιων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έγινε η μεγάλη διεύρυνση το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένταξη μεγάλου αριθμού νέων χωρών μελών, στη Γερμανία είχαμε τότε σοσιαλιστές στην κυβέρνηση και αριστερά και η Γερμανία δεν ήταν από τις χώρες που τάχθηκαν υπέρ μιας ανοιχτής πολιτικής ελεύθερης διακίνησης ε, των πολιτών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά περιόρισαν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οπότε η προάσπιση των συνόρων, της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ε, ε, συνοχής για μια χώρα είναι πολύ θεμητή προσπάθεια. Και Επίσης, αν δημιουργούμε φρούδες ελπίδες στους πρόσφυγες και μετανάστες, νομίζω ότι τελικά το κακό τους θα επιτύχουμε. Γιατί έτσι θα, δώσουμε, ε, θα αφήσουμε ανοιχτό το δρόμο και στην παράτυπη μετανάστευση με τις γνωστές τραγικές συνέπειες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τα αίτια για τις μεταναστευτικές διαδρομές, αλλά να σεβαστούμε την εθνική κυριαρχία ε, και από άποψη νομική και από άποψη αξιών. Μόνο τότε, περιλαμβάνοντας και αυτές τις θεωρήσεις, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Επίσης, ε, Υπάρχει πολύ διαφορετική εντύπωση για την οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και εδώ υπάρχουν διαφορές. Εμείς τουλάχιστον σεβόμαστε την αρχή της μονογαμικής οικογένεια, ενώ οι μουσουλμανικέ χώρες από, την, από το Μαρόκο μέχρι την Ινδονησία έχουν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της οικογένεια γιατί εκεί ισχύει πολυγαμία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Γιουρέκ και το λόγο έχει ο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για το κάλεσμα των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε σημερινή σας συζήτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχθεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων από διάφορε χώρε τη Ασία και τη Αφρική. Οι άνθρωποι αυτοί πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα είτε να παραμείνουν για ένα μακρό χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε να εγκατασταθούν μόνιμα στα κράτη-μέλη τη. Επομένω, ή όσο το δυνατόν ταχύτερη και πληρέστερη ενσωμάτωσή του στι τοπικέ κοινωνίε και την αγορά εργασία αποτελεί υψίστη προτεραιότητα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να στήσουν από την αρχή τι ζωέ του και να μπορέσουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αυτοσυντηρηθούν. Και πάντα μιλάμε κυρίω για πρόσφυγε και για νόμιμου μετανάστε. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δραστική μείωση του χρόνου εξέτασης των, ετοιμών, των ασύλου, ώστε να διευκρινίζεται άμεσα το νομικό καθεστώς όσων πράγματι μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες. Από τη στιγμή που αυτό θα διευκρινιστεί, τα δύο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν <clears throat> είναι η κοινωνική ένταξη και η εξέβρεση θέσεων εργασίας για τους πρόσφυγες. Πρόκειται προφανώς για δύο διαδικασίες που είναι απολύτω αλληλοεξαρτώμενες. Η πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς οργανωμένο σχέδιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε να εγκατασταθούν σε περιοχές που μπορούν όντως να βρουν δουλειά. Μια δουλειά η οποία ταιριάζει με τις δεξιότητες που διαθέτουν. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων είναι προς το συμφέρον τόσο των προσφύγων όσο και των κρατών υποδοχής. Παράλληλα οφείλουν να υπάρξουν πρόνοιες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξοικείωση των προσφύγων με την τοπική γλώσσα, ώστε να υπάρχει μια επικοινωνία. Δίχως την εξασφάλιση της γλωσσικής επάρκειας, το επαγγελματικό μέλλον των προσφύγων θα είναι αμφίβολο. Η εξέβραση εργασίας αποτελεί ασφαλώς το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων. Όσο, όσο οι πρόσφυγες εξαρτούνται από την κρατική ή άλλη βοήθεια για την επιβίωσή τους, τόσο θα τείνουν να περιοθεροποιούνται σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα, η οικονομική ανεξαρτοποίησή τους αφενός θα τους επιτρέψει να σταθούν μόνοι στα πόδια τους και αφετέρου θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αποδυτικότερη όσμωσή τους με τις τοπικές κοινωνίες. Ω προ την τοπική ένταξη καθοριστική ασφαλώς είναι η πρόσβαση των παιδιών σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των προσφύγων σε υπηρεσίες υγείας. Πολύ σημαντική επίσης είναι η διευκόλυνση των προσφύγων στην εξέβρεση αξιοπρεπών κατοικιών. Οι αποτελεσματικέ πολιτικέ κοινωνική ένταξη δεν μπορεί παρά να ενθαρρύνουν την όσβαση των προσφύγων με τι τοπικέ κοινωνίε και να αποτρέψουν τη δημιουργία συνθήκων διαχωρισμού των προσφύγων. Ωστόσο, θα πρέπει εξίσου να λαμβάνεται υπόψη αφενό οι τοπικέ ιδιαιτερότητε των κρατών υποδοχή. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένω από του έγκριτους κυρίου βουλευτέ. Εθνική, γλωσσική, θρησκευτική, οι ιδιαιτερότητε οι οποίε θα υπάρχουν και επικοινομορφία των προσφύγων. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στι ιδιαίτερε συνθήκε που επικρατούν σε κάθε περίπτωση. Σε όλε αυτέ τι διαδικασίε, ο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι καθοριστική σημασία. Εκείνοι του υποδέχονται. Εκείνοι του έχουν και, και ζουν μαζί του. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ είναι εκείνε που πρώτε από όλε καλούνται να αντιμετωπίσουν επιτόπου μόνο την αρχική περίθαλψη αλλά και τελικά και την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των προσφύγων. Σε τελική ανάλυση, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ είναι αυτέ που θα διαχειριστούν στην πράξη τόσο την επαγγελματική όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων. Καμία εθνική ή ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα πετύχει αν δεν έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντα υπόψη τι απόψει των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η ενσωμάτωση των προσφύγων είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει χρόνια. Χρειάζεται σχέδιο και αποφασιστικότητα. Η πείρα των τελευταίων αυτών έχει αποδείξει στην πράξη ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι οι φορείς εκείνοι που μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο της προσφυγικής ένταξης. Γι' αυτό το λόγο οι εθνικές κυβερνήσεις και πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την όποια αλλά αναγκαία βοήθεια στι τοπικέ και ευρωπαϊκές αρχέ, προκειμένου να φέρουν ει πέρα αυτήν την εξαιρετική και σημαντική αποστολή του. Επίση, θα ήθελα να προσθέσω το εξή και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνεργασία με τι τοπικέ και περιφερειακές αρχές, έτσι ώστε η συμβολή του να είναι ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική και αφετέρου να είναι συμβατή με τι τοπικέ ανάγκε και συνθήκε, Αλλά και θα πρέπει, και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, να υπόκεινται στην απαραίτητη κοινωνική λογοδοσία. Πού πήγαν τα χρήματα, τι το που πιάσανε και τι έγινε. Θα θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι οι δήμαρχοι και κυρίως οι δήμαρχοι του Αιγαίου, των νησιωτικής ζητούν περισσότερο βοήθεια ώστε το άσυλο να δίνεται εντός δύο μηνών προκειμένου να ξεχωρίζουν οι διαδικασίες αυτές. υπεύθυνο στο hot spots που είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι στη Μυτιλίνη που μίλησε ο συμπατριώτης μου ο βουλευτής προσέξτε ο Μοριάς το hot spot είναι για 3.000 άτομα και είναι 9 και 10.000 άτομα. Και αυτοί οι άνθρωποι περιφέρονται. Άρα λοιπόν εγώ κλείνοντας θέλω να σας πω ότι εμείς σκεπτόμαστε σαν τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές ότι αν η Ευρώπη, εσείς δηλαδή οι Ευρωβουλευτέ και τα Εθνικά Κοινοβούλια υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους και μπει ένας προγραμματισμός, ο λαϊκισμός δεν θα υπερισχύσει. Δεν θα είναι πρώτη ατζέντα στις ευρωπαϊκές ή τοπικές εκλογές, εθνικές, το θέμα του μετανάστη, ώστε όποιος κλείνει τα σύνορα να κερδίζει τις εκλογές. Η Ευρώπη έχει σαν επίκεντρό τη τον άνθρωπο. Και αυτό πρέπει να παραμείνει. Αυτός είναι ο πολιτισμός της, αυτή είναι η κουλτούρα της. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. We... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε δύο συναδέλφους από το Κοινοβούλιο, την Τζιν Λάμπερτ και μετά την κυρία Βερζιά και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν πριν ολοκληρώσουμε. Τζιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Είμαι εδώ εν μέρους ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και φυσικά και ως μέλος τη Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Εξετάζουμε την ε, μετανάστευση για λόγους εργασίας από διαφορετικό οπτικό πρίσμα στην Επιτροπή Απασχόλησης και νομίζω ότι το βασικό μήνυμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε από αρκετά μέρη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από αρκετά κράτη-μέλη είναι ότι ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος ε, για ένα μικρό διάστημα αλλά μετά πρέπει να αποχωρήσουν που δεν είναι απαραίτητο αυτό που επιθυμούν οι εργοδότες. Επιθυμούν ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, παραμένουν, ε, αναπτύσσονται και συμβάλλουν και με τις δεξιότητές τους και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα μόνο της παγκόσμιας μετανάστευση. Ε, δεν είμαστε ο φάρος μέρος του κόσμου και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσελκύσουμε αλλά και να διατηρήσουμε τα ταλέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε κάποια αναφορά στην μπλε κάρτα, κάποια από τα ερωτήματα στο θέμα αυτό αφορούν και την επανόνωση των οικογενειών, ε, ε, ο κόσμος θέλει να έρθει, υπάρχουν οι λεγόμενοι σύζυγοι και σύντροφοι που θέλουν να έρθουν αλλά και να εργαστούν. Ε, δεν ε, είναι ικανοποιημένες οι γυναίκες να κάθονται στο σπίτι και να κεντάνε. Ε, και φυσικά η κάθε χώρα έχει διαφορετικό ορισμό της οικογένειας. Αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε είναι ότι γνωρίζουμε τι απαιτούμε από τους ανθρώπους που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε αρκετά από αυτά σήμερα το απόγευμα, αλλά το θέμα είναι τι τους προσφέρουμε αν πραγματικά θέλουμε να αποτελέσουμε και δέλεαρ, γιατί ακούστηκε και σε μια διάσκεψη που έκανε η Εστονική Προεδρία, ότι δεν ανοίγουμε απλώς την πόρτα, πρέπει να ζεστάνουμε και το σπίτι για να τους υποδεχθούμε. Τι προσφέρουμε λοιπόν ε, το οποίο ε, θα προσελκύσει ε, νέους ταλαντούχους ανθρώπους με δεξιότητες για να έρθουν εδώ όταν ακούν τον τρόπο με τον οποίο συζητούμε τη μετανάστευση. Αποτελούμε εμείς δέλεαρ. Ευχαριστώ, Τζίνι, Μαρή Κριστίν Βερζιά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ από πλευρά μου είμαι μέλο τη Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ και τη Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και είμαι και η ε, εισηγήτρια μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν συζητούμε αυτά τα θέματα, αυτό το οποίο που με ενδιαφέρει να τα θέσουμε στο ιστορικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο και όταν ακούμε τις διάφορες απόψεις, δίνεται εντύπωση ότι δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα όταν αναφερόμαστε στους μετανάστες. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αν δούμε τα στοιχεία χονδρικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η, μέση, η ε, μισή μετανάστες είναι περίπου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι μία από τις μεγάλες ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι και να λέμε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Σέγγεν, θα μπορούσε ίσως ε, να είναι εις βάρος αυτής της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, και ε, να είναι εις βάρος και των χωρών ε, Ανατολών. Μιλάμε για τους μετανάστευς, λες και δεν υπάρχει πλέον νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, δίνουν πάνω από 3 εκατομμύρια άδειων παραμονής και διαμονής. Δεν ξέρω ακριβώς τα ακριβή στοιχεία, μισό λεπτό κάπου εδώ τα είχα. Για για πέρσι, για το 2016, είχαμε 3.400.000. Δεν έχω ακόμα τα στοιχεία του 2017. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός, ε, ιδιαίτερα από το 2012 και μετά, ε, και το 2012 ήταν η χρονιά με τις ε, λιγότερες αφήξεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη συμπεριφέρονται με τελείως διαφορετικό τρόπο όσον αφορά αυτές τις άδειες παραμονής, που είναι ουσιαστικά η νόμιμη οδός μετανάστευσης. Η το πρώτο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το Brexit. Ε, κάθε χρόνο δίνει 800.000 άδειε παραμονής, ε, κυρίως ε, Κινέζοι, Ινδοί και από τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι αυτοί που έρχονται. Και επίσης η Πολωνία είναι αυτή η οποία δίνει πολύ μεγάλο αριθμό επίσης αδειών παραμονής και το 80% αυτών των αδειών παραμονής είναι άδειε εργασίας για να μπορούν να έρθουν Ουκρανοί να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως υπάρχει οικονομική μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμένα με εκπλήσει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις πολιτικές των κρατών μελών για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Και αυτό φυσικά ε, γίνεται αντιληπτό αν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Ε, Κάποιο Γάλλος ε, κοιτάμε τις παλιές απικίες εντό εισαγωγικών ε, όταν κάποιος είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συγκεκριμένες συμφωνίες με, χώρες, με τις χώρες της κοινοπολιτείας και φυσικά στην Ανατολή, στην Πολωνία ε, στρεφόμαστε προς την Ουκρανία. Ε, δεν υπάρχει βέβαια λόγος να ομογενοποιηθούν οι κανόνες αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την κατάσταση συνολικά και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σωστά για τα πράγματα και να δώσουμε σαφή στοιχεία. Γι' αυτό το οποίο με εκπλήσει όταν συζητάμε για τους μετανάστες και κάνουμε την παράλογη διαφοροποίηση μεταξύ πρόσφυγα και ε, οικονομικού μετανάστη, ε, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες ε, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να έχουν νόμιμες οδούς για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι άλλους για τους οποίους δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες διευκόλυνσης. Εάν προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις χώρες, τι γίνεται με το σύστημα απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα να δούμε την πραγματικότητα και όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και τελευταία σύντομη παρέμβαση πριν περάσουμε στο πάνελ των καλεσμένων μας. Κύριε Βότσεχα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ως μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διαπιστώνουμε σήμερα τι ε, διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΜΕ θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενσωμάτωσης και προσφύγων. Αφού το ακούσαμε ξεκάθαρα σήμερα. Κάποιοι θέλουν ε, οι πρόσφυγες ε, να μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται την γλώσσα, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Έχει δίκιο βέβαια και ο κύριος Μάιερ που μίλησε για τη συνθήκη της Γενέβης και την υποχρέωση που προκύπτει από αυτή. ότι όταν ε, πάυσει η αιτία για την οποία έφυγαν οι πρόσφυγες ε, μα ε, πρέπει να επιστραφούν και γιατί λοιπόν στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η ενσωμάτωση και υπάρχει λοιπόν αυτή η διάκριση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της ενσωμάτωσης και των προσφύγων αλλά ως τώρα Δεν υπάρχει επαρκή συνδιάκριση, θεωρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των πρόθυμων και των απρόθυμων. Πώς να ενσωματώσω κάποιον που δεν θέλει να ενσωματωθεί. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και την θρησκευτική προέλευση του πολιτισμικού κύκλου και νομίζω ότι εδώ η Πολωνία βρήκεται στην σωστή κατεύθυνση γιατί οι Ουκρανοί προφανώς και συγκαταλέγονται στη χριστιανική δύση. Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, σήμερα κάνουμε σήμερα αυτό που δεν κάνανε τα τελευταία 100 χρόνια οι επικοινωνικές δυνάμεις της Ευρώπης. Αυτό όμως είναι άλλη ιστορία. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κουρτέ, έχει το λόγο για να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πολλά σχόλια, πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να επανέλθω σε μερικά από τα σχόλια γιατί όλα αποκλείεται. Θα χρειαζόταν να μακρηγορήσω. Κάτι που αναφέρθηκε ιδιαίτερος είναι η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Το διεθνές δίκαιο τουλάχιστον προβλέπει διαφορετικές υποχρεώσεις για τα κρατημέλη ανάλογα με το αν πρόκειται για πρόσφυγα ή για μετανάστη. Σε περίπτωση των προσφύγων έχουμε ανθρωπιστικά ζητήματα, ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους ε, λόγω ανασφάλειας, ε, έλλειψη ασφάλειας μάλλον, σύραξης, ε, πολέμου, δίωξης και υπάγονται στη συνθήκη της Γενέβης με αρμόδια την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Το θέμα, η για μεταναστη σε περιπτωση των προσφυγων εχουμε ανθρωπιστικα ζητηματα ανθρωπων που εγκαταλειπουν τη χωρα τους λογω ανασφαλεια ελλειψη ασφαλεια μαλλον συραξη πολεμου διωξη και υπαγονται στη συνθηκη τη γενεβη με αρμοδια την υπατη αρμοστια των ηνωμενων εθνων το θεμα η περιπτωση του μετανάστη είναι διαφορετική και γι' αυτό οι πρόσφατες εξελίξεις στα Ηνωμένα Έθνη προέβησαν και σε αυτή τη διάκριση. Ε, ακούσατε το πρωί για τα δύο σύμφωνα που επεξεργάζονται τα Ηνωμένα Έθνη. Το ένα σύμφωνο αφορά τους πρόσφυγες και το άλλο σύμφωνο αφορά τους μετανάστες. Και ακριβώς αυτό έγινε για να καλυφθούν οι διαφορετικές περιστάσεις και τα διαφορετικά ζητήματα. Όπως είπα στην δική μου ομιλία, η μετανάστευση θα πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και αυτό συνάδει με τα σχόλια της Ομίγυρης ε, ε, για το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης ή όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το επιχείρημα ε, που υπερισχύει είναι αυτό που, θα, είναι αυτό που συνδέει τη μετανάστευση, την οικονομική μετανάστευση με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Και αν σκεφτούμε τις πρόσφατε εμπειρίες μα ε, και προσπαθήσουμε να ταινίσουμε και το μέλλον, αυτή η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών ίσω σε μερικέ περιπτώσει γίνεται ασαφή και ρευστή. Το ζήτημα αυτό το ε, πραγματεύεται και ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην τελευταία του έκθεση. Υπάρχουν όλο και περισσότερε περιπτώσει που άνθρωποι ξεριζώνονται, όχι κατά ανάγκη λόγω του πολέμου, αλλά εξαιτία τη δινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν στη χώρα του. Ένα από τα ζητήματα που εξετάστηκε και συζητήθηκε ευρέω τουλάχιστον στα Ηνωμένα Έθνη είναι το θέμα των περιβαλλοντικών προσφύγων ή κλιματικών προσφύγων. Και ιδιαίτερα άνθρωποι που διαβιούν στην υποσαχάριο Αφρική και που η επιβίωσή τους συνδέεται με τη γη τους, όταν υπάρχει ξηρασία, παρατεταμένη ανοβρία, δεν μπορούν πια να επιβιώσουν. Αυτοί είναι πρόσφυγες λόγω, μετανάστες λόγω κλιματικών αλλαγών. Η κατάσταση λοιπόν μερικές φορές είναι σαφής και ρευστή μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. Ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που μετα, μετακινούνται αναγκαστικά όμως, δεν έχουν επιλογή. Ένα άλλο ε, θέμα συνδυάζεται με αυτό που είπε ο Γερμανός ε, ε, βουλευτής για την ανάγκη αρρωγής της χώρας προέλευσης και την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης. Γιατί όσοι εγκαταλείπουν τις χώρες τους αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες, γιατί δεν έχουν αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες ή ευκαιρίες εργασιακές στην πατρίδα τους. Και ε, ξεριζώνονται αναζητώντα ένα καλύτερο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να ε, αντιμετωπίσουμε τα αίτια τη μετανάστευση, ώστε ο κόσμο να παραμένει στην πατρίδα του και να μπορεί να επιβιώνει, όχι σε άθλιε συνθήκε. Ξέλιφοντα δηλαδή τη φτώχεια. Επίση, ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τι αφρικανικέ και ασιατικέ χώρε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στι χώρε αυτέ. Επίση, υπάρχει το πρόβλημα τη διαφυγή των εγκεφάλων τη απώλεια ε, μετακίνηση των δεξιοτήτων. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε μια χώρα, δεν γίνεται αν όλο το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχει ήδη αποδημήσει. Για τον τομέα της Υγεία είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν αφρικανικέ χώρε που έχουν μείνει χωρί γιατρού, χωρί νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όλε οι νοσοκόμε, όλοι οι νοσηλευτέ και οι γιατροί έχουν αποδημήσει την Ευρώπη. Οπότε ε, έχουμε ενδιαφέρουσες ε, εμπειρίες προσπαθώντας να αντικαταστήσουμε τη διαρροή εγκεφάλων με την προσέλκυση εγκεφάλων, ώστε να έχουμε μια υποφελή λύση για όλες τις πλευρές και να ε, αξιοποιήσουν όλοι τις δεξιότητες των εργαζομένων. Αυτό είναι σημαντικό πάντω για τι αναπτυσσόμενε χώρε να μην έχουν τέτοια διαρροή εγκεφάλων. Αναφέρθηκε το θέμα τη εμπορία ανθρώπων ή τη λαθροδιακίνηση. Σα ευχαριστώ που το θίξατε γιατί δυστυχώ είναι πραγματικότητα στην Ευρώπη. Έχουμε την τάση να, σκεφτόμαστε ότι η αναγκαστική εργασία ή η εμπορία ανθρώπων ή ε, μεγάλη εκμετάλλευση δεν υπάρχει, αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί στη ΔΟ έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και από κοινοτικέ χώρες που εντοπίστηκαν τέτοια φαινόμενα υπάρχει ο κίνδυνος της ε, εργασιακής εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκμετάλλευση από τον εργοδότη τους. Αυτό που είπα στην ε, ομιλία μου και πολύ ευχαρίστω να παραμείνω για να το συζητήσουμε πιο δεξιωτικά αργότερα, είναι σημαντικό να έχουμε ίση ε, μεταχείριση, που φυσικά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν ισχύει πάντα, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το στόχο και να ενισχύσουμε τους φορείς εργασιακής επιθεώρησης, με συνεργασία με τις ομάδες ε, της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικέ κυβερνητικές οργανώσεις, ε, συνδικάτα και ομάδες εργοδοτών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους που εντοπίζονται περισσότερο αυτά τα φαινόμενα της εκμετάλλευσης. Και τέλος, ε, σε σχέση με αυτά που ρώτησε η Τζιν, τι θα προσφέρουμε στους ταλαντούχους νέους που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Θα ήθελα να δώσω μια γενική απάντηση άσχετα πρόκειται για ταλαντούχους ε, υπερειδικευμένους ή ανειδίκευτους ή χαμηλά ειδικευμένους, αν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και θέλουμε η ανειδικευτου η χαμηλα ειδικευμενου αν οικονομία να γίνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το δυναμικό, σε αυτές τις δεξιότητες, στην εκπαίδευση. Και όταν να επενδυσουμε σε αυτο το δυναμικο σε αυτε τι δεξιοτητε στην εκπαιδευση και οταν λεω επενδυση δεν είναι μια λέξη που διαλέγω τυχαία. Δεν πρόκειται για κόστο, δεν πρόκειται για δαπάνη, αλλά για επένδυση και θα πρέπει να αφιερώσουμε αυτά τα κονδύλια, αυτέ τι επενδύσει, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα. Και φυσικά θα υπάρξουν και δημοσιονομικέ συνέπειε. Δεν θα γίνεται κάτι τέτοιο δωρεάν. Δεν θα προσελκύουμε αυτού του ανθρώπου, θα του χρησιμοποιούμε στην οικονομία μα. Πρέπει να επενδύσουμε και στην κατάρτισή του, στην παιδεία του, στην επιμόρφωσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ συχνά η οικογενειακή επανένωση δεν ε, γίνεται σωστά αντιληπτή. Και εσείς ε, που πρωτοστατείτε στη δημόσια συζήτηση θα πρέπει να μιλήσετε για τους πρόσφυγες και τους ε, μετανάστες ως μέλη οικογένειας και να ασχολήσετε και με τις οικογένειές τους και να τονίζετε τα δεινά που υφίστανται. Γιατί πολύ συχνά εξετάζουμε τα νούμερα και νομίζουμε ότι σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Η οικογενειακή επανένωση είναι ο καλύτερο διάβλος που έχουμε για ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση. Γιατί πολλές χώρες προσπαθούν να επινοήσουν νέα προγράμματα, νέα συστήματα, επανεγκατάσταση, υποτροφίες για πρόσφυγες και υπάρχουν τέτοια χορηγούμενα προγράμματα, επιχορηγούμενα, αλλά η οικογενειακή επανένωση είναι αυτή που επιτρέπει στις συζύγους, στα τέκνα να ε, επανενωθούν με τον σύντροφο που έκανε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη. Αυτό είναι το θεσμοθετημένο σύστημα, το μοναδικό θεσμοθετημένο σύστημα που έχουμε με ε, τις οικογένειες που εγκαθίστανται τοπικά, με μια, νέα ασφαλή, με μια νέα ασφαλή αιστεία, τα παιδιά να σπουδάζουν στα τοπικά σχολεία και με ε, χρόνο για να εξεταστεί η αίτησή τους και η διαφορά με το σύστημα επανεγκατάστασή τους αυθόρμετους αυθόρμητα του άσυλο ε, δεν είναι μια σωστή διάκριση, σωστός παραλληλισμό, Όσοι ε, μπορούν να, ανατύχουν τη της οικογενειακής επανένωσης ε, μάλλον θα μείνουν πολύ περισσότερο καιρό στη χώρα. Και μάλιστα οι μακροχρόνιες επανεγκαταστάσεις μεταναστών βελτιώνει την την κοινή αντίληψη για το μεταναστευτικό φαινόμενο. Και σίγουρα η οικογενειακή επανένωση είναι σημαντικός συντελεστής που συμβάλλει αρνητικά όταν καθυστερεί και δημιουργεί δευτερογενείς κινήσεις και έχει και αρνητικά αποτελέσματα μια τέτοια καθυστέρηση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στις διαδικασίες ενσωμάτωσης κοινωνικής ένταξης και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η μέση σύραξη ε, διαρκεί πια μια δεκαπενταετία. Δεν μιλούμε για ένα εφήμερο φαινόμενο, για μια προσωρινή πραγματικότητα. Και στη Γερμανία οι περισσότεροι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας που άσκησαν προσφυγή στην απόφαση κέρδισαν το ένδικο μέσο και τελικά απέκτησαν καθεστώς πρόσφυγα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε με κριτικό μάτι τις πολιτικές οικογενειακής επανένωσης και να διαπιστώσουμε ότι μέχρι στιγμής κάνουν το βίο αβίωτο, τον οικογενειακό βίο αβίωτο αυτών των ανθρώπων. Μερικές φορές α, τη ζωή τους μόνο και μόνο για να συνδεθούμε με την οικογένειά τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε άλλους κανόνες, μια ε, περιπτωσιολογική ανάλυση καλύτερα και αν θέλετε περισσότερα στοιχεία για την καλύτερη λειτουργία των πολιτικών ε, οικογενειακής επανένωσης, καλύτερα μιλήστε με οργανώσεις ε, προστασίας των οικογενειών στις πατρίδες σας. Αυτές γνωρίζουν πολύ καλύτερα για το πώς ε, βοηθούν τις οικογένειες και είναι υπέρ της διευκόλυνσης της οικογενειακής επανένωσης. Και θέλετε περισσότερα στοιχεία για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις πολιτικές ένταξης για ενήλικες ε, και γυναίκες. Μιλήστε με τον, την υπατερμοστία τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως για την ένταξη των παιδιών. να έρθετε σε επαφή με το δίκτυο πολιτικής ε, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δεν χρειαζόμαστε νομικές νομοθετικές αλλαγές, χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και καλύτερη στήριξη της κοινωνικής ένταξης από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα που θα εφαρμόζονται όμως εμπράκτος από τα κράτη-μέλη, τις κεντρικές και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που έλαβαν το λόγο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που δεν αναφέρθηκε ακόμη. Θα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ε, έναν έλεγχο καταλληλότητας ε, και αξιολόγησης και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί θέλουμε ε, να δούμε πώς ε, ε, νομοθεσία που ισχύει εδώ και δεκαετία εφαρμόζεται στην πράξη και αν εφαρμόζεται σωστά. Και θα ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα συμπεράσματά της από, την, από τον έλεγχο αυτών της καταλληλότητας και ποιες είναι οι συστάσεις της για το μέλλον. Και μετά τους νόμους διάβλους και το θέμα το πώς θα εξασφαλίσουμε ε, οι Τρίτοι χωρών που φτάνουν, ε, να φτάνουν στο, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς οι αφιχθέντες μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στις νέες κοινότητες. Για να τα ακούσουμε όλα αυτά θα δώσω το λόγο στην Τζέιν Λάμπερτ, την εξαιρετική συνάδελφο και εισηγήτρια της ε, Επιτροπής Απασχόλησης για την Οδηγία για την Μπλε Κάρτα, έχει όμως προωθήσει και παρακολουθήσει πολλά ζητήματα ασύλου και μετανάστευση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών πολύ πήρε ευρωβουλευτής, ε, μακροχρόνια θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σίγουρα θα σας καθοδηγήσει επιδέξια στην επόμενη φάση της συζήτησης. Okay, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε και πάλι. Γιατί όσο καθυστερήσουμε, τόσο λιγότερο χρόνο θα έχουμε για τη συζήτηση. Γιατί φυσικά και, και εσείς έχετε τα τρένα σας, έχετε τα αεροπλάνα σας και το χρονοδιαγραμμά σας. Η συνάδελφος, η κυρία Μετσόλα, ε, σας είπε ότι είμαι η Τζιν Λάμπερτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια. Όπως είπα και προηγουμένως, είμαι μέλος και της Επιτροπής Επασχόλησης και της Επιτροπής ε, για τα Δικαιώματα του Πολίτη. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη συνεδρία για τα θέματα που άπτοντα της ε, ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, ευκαιρίες ε, και προκλήσεις. Θα εστιαστούμε λοιπόν στην ενσωμάτωση υπηκόνων των χωρών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός κράτους, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι οικονομικοί μετανάστες. Και νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθνικών, με τις εθνικές, με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί είναι πολλές και κοινέ οι αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών και στο ιστορικό των κρατών μελών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κυρίως εστιάζονται οι δράσεις για την ενσωμάτωση των προσφύγων. Άρα, θα ακολουθήσουμε την εξή ε, σειρά. Καταρχάς, θα ακούσουμε τα αριθμητικά στοιχεία και τα πρόσφατα απορίσματα σε ό,τι αφορά τις πρακτικές ενσωμάτωσης ε, βάσει μέλετων του ΑΣΑ και των, του... των υπηρεσιών θεμελιδιών δικαιωμάτων. Ο κ. Λίμπη και ο κ. Παύλου θα είναι υπεύθυνοι για την παρουσίαση των στοιχείων αυτών. Μετά θα ακούσουμε συγκεκριμένες εμπειρίες ε, από τον κύριο Κίμιλο, ο οποίος είναι γερμανός επιχειρηματίας με μα, προέλευση πρόσφυγα και ο ίδιος, μεταναστευτική μάλλον ε, προέλευση. Μετά θα ακούσουμε την κυρία Αρμαντόρ που θα μας μιλήσει για την κατάσταση στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και θα ακούσουμε επίσης τον κύριο Δημήτριο Κάλο Γερόπουλο από την Επιτροπή των Περιφερειών. Και μετά θα έχουμε μια συζήτηση. Πρωτού, ωστόσο, ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι μοντέλα ακολουθούμε για τη συζήτηση. Θα δώσουμε το λόγο σε δύο μέλη του Αθηνικών Κοινοβουλίων και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Τα μέλη των Αθηνικών Κοινοβουλίων, ε, αν επιθυμούν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ να συμπληρώσουν το έντυπο αυτό, το κίτρινο έντυπο για την απογευματινή συνεδρία και να δώσουν το έντυπο αυτό στην γραμματεία. Α, όχι μπλε, μάλιστα, πολύ ωραία. Μετά λοιπόν θα καταφθήσουμε το μετάλλαγμα των ομιλητών με τη σειρά που θα λάβουμε τα φυλάδια και οι βουλευτές παρακαλώ να επισημάνουν ευγενικά ότι επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Και ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα θέλουν να πάρουν το λόγο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εξίσου αυστηροί με το χρόνο ομιλίας. Τουλάχιστον δύο λεπτά όμως θα σας ε, δώσουμε. Είμαστε πολύ γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά το χρόνο ομιλίας. Εκτός βέβαια και αν ε, είναι κανείς μέλος του Προεδρείου, στην οποία περίπτωση μπορεί να μιλήσει ο θέλει, όπως κάνω και εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Λίμπεκ από τον ΩΣΑ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που μας κάλεσε για να παρουσιάσουμε το έργο μας. Θα επικεντρωθώ κυρίως στην αγορά εργασία ό,τι αφορά την ενσωμάτωση. Γιατί η ενσωμάτωση στην αγορά εργασία, όπω ξέρουμε, είναι το ένα και μοναδικό πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να πετύχουμε για να υπάρχει αυτή η ευκταία ενσωμάτωση στην κοινωνία. Αυτό άλλωστε εμ, επιθυμούμε όλοι και οι μετανάστε, ε, Τι σημαίνει για το μετανάστη να ενσωματωθεί, να είναι ανεξάρτητο και να βρει δουλειά. Βλέπετε κάποια απορίσματα από έρευνες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την ε, κρίση την προσφυγική και κάναμε και κάποια ανάλυση με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης. Και βλέπετε λοιπόν δύο πράγματα. Καταρχάς ότι η ενσωματώση είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Χρόνο και γενικώ τα αποτελέσματα βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Και κατά δεύτερον βλέπετε ότι εξαρτάται ε, από το ποια κατηγορία, σε ποια κατηγορία υπάγεται κανείς. Και ότι είναι σημαντικό, όπω είπατε, να κάνουμε αυτή την κατηγοριοποίηση των μεταναστών, γιατί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά και την αγορά εργασία. Βλέπετε πώ ε, είναι η πορεία για την απασχόληση χαμηλά ποσοστά στην αρχή και μετά πρόοδο. Αλλά και πάλι παίρνει 15 χρόνια μέχρι ότου να φτάσουν σε μια παρόμοια κατάσταση εργασιακή με τον αυτόχθονα πληθυσμό. Οι μετανάστες θα πηγαίνουν κάπως καλύτερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι κυρίως γυναίκες. Κοιτώντα τώρα τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφορά τα πορίσματα και κοιτάξουμε του πιο Χαμηλή εκπαίδευση ε, εργαζομένου. Βλέπετε λοιπόν του Χαμηλή εκπαίδευση, ότι είναι αρνητικό, το κάνω λιγότερο, ότι είναι θετικό, το κάνουν πιο καλά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι μισές χώρες του ΟΣΑ οι χαμηλή εκπαίδευση μετανάστε τα πηγαίνουν εξίσου καλά με του υπόλοιπου υψηλή εξειδικεύση. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται στι χώρε που τα πηγαίνουν άσχημα σχετικά. Τα πηγαίνουν άσχημα όχι για την απαραίτητα κακή πολιτική ενσωμάτωση, αλλά έχουν ε, δεχτεί κατηγορίε που αντιμετωπίζουν πιο πολλέ δυσκολίε. Αυτό είναι στοιχεία πριν από την μεταναστευτική κρίση, από την προσφυγική κρίση. Ενημερώνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τις, ε, λίστες στους καταλογούς αυτούς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Προετοιμάζουμε την έκδοση του 2018, την οποία με χαρά θα σας ε, χορηγήσουμε όταν ε, ετοιμαστεί. Άρα έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά πολλούς πρόσφυγες που τα πηγαίνουν ε, μάλλον άσχημα και έχουμε χώρες που έχουμε χαμηλής εξειδίκευσης μετανάστευση, όπως ήταν για παράδειγμα χώρες της Νότιας Ευρώπης πριν από την οικονομική και προσφυγική κρίση. Αλλά αυτό εξακολουθεί να ισχύει για παράδειγμα και στη ΣΥΠΑ. Εκεί οι μετανάστες τα πηγαίνουν καλύτερα από τις χαμηλές εξειδικεύσεις, ε, χαμηλές εκπαιδευσής ε, αυτόχθονες. Όταν βλέπουμε λοιπόν όμως τι γίνεται στα άτομα υψηλής εξειδικεύσης, εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα παντού και στις χώρες χρυσών ευκαιριών όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία που γενικά αποτελούν καλά παράδειγματα. Εκεί πέρα λοιπόν ακόμα και εκεί τα άτομα υψηλή εξειδίκευση ε, και ψηλή εκπαιδευτικού επίπεδου τα πηγαίνουν χειρότερα. Και έτσι λοιπόν ε, μιλάμε για μια κατάσταση όχι win-win, αλλά lose-lose, όχι αμοιβαία αποφελή, αλλά αμοιβαία αρνητική, γιατί χάνει και η χώρα που χάνει τους υψηλής εκπαιδευτείς και εξειδικευσής ε, εργαζόμενους και η χώρα η οποία τους υποδέχεται. Αυτό είναι πιο, πολύ πιο συνήθες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε τους ε, μετανάστες ό,τι αφορά τις δεξιότητες. Ξεκινάμε εντοπίζοντας τις δεξιότητες που έχει ο κάθε και στη συνέχεια αντιπιστώνουμε ότι προφανώς κάποιοι πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες. Η πιο προφανής είναι η γλωσσική δεξιότητα, αλλά και άλλα ζητήματα. Και πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν περαιτέρω κάποιε ικανότητε, δεξιότητε. Στο τρίτο τμήμα λοιπόν έχουμε την δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση των δεξιοτήτων για να χρησιμοποιηθούν επαρκώ στην αγορά εργασία. Μεταφορά λοιπόν ε, γνώσεων για την λειτουργία της αγοράς εργασίας και το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης προφανώς είναι σημαντικό στο σημείο αυτό. Σε επίπεδο ωσα με το Υπουργείο Εργασία της Γερμανίας και το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, κάναμε μια μελέτη ε, σε 2.000 Γερμανούς εργοδότες. Ρωτήσαμε λοιπόν ποια είναι η εμπειρία με τους, με τους μετανάστες ως εργαζόμενους. Και εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε κάποιες από τις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι εργοδότε. Σαφώς η γλώσσα αποτελεί το υπαριθμό ένα εμπόδιο. Έχουμε ανεπαρκείς επαγγελματικέ δεξιότητε ε, και αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το διάστημα που θα παρέμεναν. Αυτό λοιπόν αφορούσε πολλού τέτοιου εργαζόμενου και προφανώ εμποδίζει την απασχόλησή του. Αλλά 85% των ε, εργοδοτών είχαν πάρα πολύ λίγε δυσκολίε με του εργο... με και πάνω από 85% ήταν πολύ ικανοποιημένοι με του εργαζόμενου μετανάστε, γιατί θεωρούσαν ότι είχαν πολύ ε, μεγάλο βαθμό προθυμία. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε Καταρχά Καταρχά, η επαγγελματική γλωσσική κατάρτιση. Υπάρχει γλωσσική δεξιότητα και η γλωσσική εκπαίδευση. Κάθε χώρα δεν είναι μια γλωσσική εκπαίδευση. Αυτό που λείπει όμω είναι η επαγγελματική γλωσσική ε, ικανότητα. Γιατί αν θέλουμε να μπορεί να δουλέψει ο μετανάστης, θα πρέπει οι γλωσσικέ ικανότητε να ανταποκρίνονται στι ανάγκε τη αγορά εργασία. Η νομική βεβαιότητα αναφέρθηκε προηγουμένω πάρα πολύ σημαντική και αυτή σε ό,τι αφορά και εμά και σε ό,τι αφορά επίσης ε, τις δεξιότητες και τη διαρκή εκπαίδευση και ένα διαρκές ε, ε, μόνιμο άτομο σημείο επαφή σε περίπτωση που παρουσιάσουν προβλήματα. Έχουμε ένα πλήρη κατάλογο καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών και όπως είπε ο συνάδελφος μου, ο Τόμας Χαρλίσον, έχουμε και μια δημοσίευση για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των οικογενειών που περιλαμβάνει διάφορα καλά στοιχεία. Δεν θα μπω σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια, αλλά θα πρέπει ε, νωρί να εντοπιστούν οι δεξιότητε. Και όταν ξέρουμε πλέον ότι το άτομο αυτό πρόκειται να μείνει, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξη. Και ξέρουμε ότι ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης της επιτυχίας στο μέλλον, μακροπρόθεσμα, είναι αν ο, οι άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους ε, εγκαίρως όταν, ε, ιδανικά, όταν είμαστε σχετικά σίγουροι ότι θα λάβουν μια θετική απάντηση για την παραμονή της στη χώρα. Και φυσικά έχουμε και το θέμα της διαφοροποίησης ε, ανάλογα με το διάφορο επίπεδο δεξιοτήτων. Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για την ενσωμάτωση και την ένταξη. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, κοιτώντας τις ε, προσφυγικές ε, ροές ε, στην Ευρώπη. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν δυσκολίες στη ζωή τους από την Αφρική, για παράδειγμα. Έχουν πάρα πολλές ικανότητες, αλλά επίσημη εκπαίδευση έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο, λόγω των μακροχρόνιων συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τους Σύρους, του Ιρακινούς, έχουμε μεγάλο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Έχουμε συγκεκριμένες λοιπόν ομάδες προσφύγων. Δεν μπορούμε να έχουμε μία και μόνο εφάπαξ λύση για όλους, για έναν πανεπιστημιακό καθηγητή, για παράδειγμα, και για έναν άνθρωπο που δεν έχει δυσκολίε στη ζωή του ποτέ. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμογή από την άποψη αυτή. Και πιστεύω ότι μία από τι πιο συναρπαστικέ τάσει που διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα σε χώρε όπω η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία, που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την προσφυγική κρίση, είναι ότι ανθεί το κίνημα της κοινωνίας των πολιτών και οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι επί το οποίο μπορεί να βασιστούν οι χώρες υποδοχής. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, ε, στην προσφυγική κρίση, το κράτος ήταν υπεύθυνο για όλα. Έγινε μια αξιολόγηση της ε, ενταξιακής πολιτικής της Σουηδίας. Το κράτος λοιπόν τα έκανε όλα πλέον με τους αριθμούς για τους οποίους μιλάμε των προσφύγων που έχουν καταφτάσει δεν φτάνει. Ό,τι και να κάνει το κράτο. Άρα χρειάζεται εμπλοκή τη κοινωνία των πολιτών. Και αυτό θεωρώ ότι διακρίνει τι ευρωπαϊκέ χώρε ε, από τον Καναδά, για παράδειγμα, από την Αυστραλία, από τη ΣΥΠΑ, όπου η κοινωνία των πολιτών ήταν αρκετά ενεργή σε ό,τι αφορά την ένταξη, την ενσωμάτωση των προσφύγων. Τέλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί με του εαυτού μα και να αναγνωρίσουμε, να ομολογήσουμε ότι για τους ε, Πρόσφυγε χαμηλή εξειδίκευση, ο δρόμο είναι μακρύ. Άρα, καλά θα κάνουμε να το σκεφτούμε εκ των προτέρων, να είμαστε ειλικρινεί και να έχουμε ρεαλιστικέ προσδοκίε για την ενσωμάτωση στην ε, αγορά εργασία. και να του δώσουμε τι απαραίτητε δεξιότητε, γιατί ξέρουμε από άλλε έρευνε που έχουμε διεξαγάγει μαζί με τη Γενική Διεθνή Απασχόλησης, ότι το πώς ενσωματώνονται οι γονείς έχει τεράστιο αντικτύπο για τα παιδιά. Άρα, το τι κάνουν οι γονείς έχει μεγάλο αντικτύπο και για τη δεύτερη γενιά, για τα παιδιά. Και θα πρέπει να συμπεράνουμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτή την ενσωμάτωση. Ω επένδυση, κάποιο το ανέφερε προηγουμένω. Τι σημαίνει η ενσωμάτωση ω επένδυση στον κόσμο. Νομίζω ότι σημαίνει τρία πράγματα συγκεκριμένα. Θα πρέπει να εστιαστούμε στην εμ, έγκαιρη ένταξη και ενσωμάτωση. Αυτό δεν το κάνουν απαραίτητα οι χώρε. Και επίση επικέντρωση σε έγκαιρη ενσωμάτωση ε, για τα παιδιά. Ξέρουμε ότι η καλύτερη ενσωμάτωση γίνεται στην παιδική ηλικία. Συχνά όμω τα παιδιά των μεταναστών υποεκπροσωπούνται. Εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν να, να ακολουθήσουμε πολιτικέ που ενδεχομένω να μην έχουν άμεσα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι γυναίκε προσφυγέ, την ενσωμάτωσή του ε, στην αγορά εργασία. Ε, δεν ε, θα ξε... έχει αυτό αποτελέσματα απαραίτητα οικονομικά άμεσα, αλλά θα έχει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην ενσωμάτωση. Θα πρέπει να, τέλος, να υπάρχουν πολύ πιο εξειδικευμένες λύσεις για την ε, ενσωμάτωση σε ό,τι αφορά δηλαδή τις προοπτικές ε, που έχει το κάθε άτομο για να εγκατασταθεί και να ενσωματωθεί, το οποίο προφανώς εξαρτάται και από τη χώρα προέλευσης όταν αφορά τα άτομα τα οποία χρήζουν αντίθετης προστασία. Θα βρείτε λοιπόν πολλά δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μα. Ε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και Προφανώς ως μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων είσαστε άτομα στα οποία πραγματικά θέλουμε να στείλουμε τις δημοσιεύσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λίμπικ. Και ευχαριστούμε και για την προσφορά που μας κάνατε στο τέλος. Χρήσιμο υλικό και τεκμηρίωση που ε, δεν είναι γνωστή παντού. Θα περάσουμε τώρα στον κύριο Μίλτο Παύλου που θα μας ενημερώσει για τις ε, προσπάθειες του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την πρόσκληση του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση σήμερα καταδεικνύει ότι ήρθε η ώρα να εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών με σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών αρχών της Ένωσης που συμφωνήθηκαν το 2004 υπέρ ε, και των πολιτών και κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, μετρήσιμες, να έχουν ε, προστιθέμενη αξία αξιοποιώντας το δυναμικό των ε, μεταναστών. Όπως είπαμε πολύ και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα μπορούμε να στήριξουμε την ένταξη στις ευρωπαϊκέ κοινωνίες και να αποτρέψουμε τι απειλέ στην κοινωνική συνοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω είναι η, ε, η ριζοσπαστικοποίηση, η μυσαλλοδοξία και το καθεξής. Τώρα συγκεκριμένε δράσει για την απασχόληση. Ήδη έχουμε πολλές ιδέες, ε, καλέ πρακτικέ για την έμπρακτη ε, κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Και μάλιστα είχαμε ενδιαφέροντα στοιχεία από τον Τόμας Λίμπικ ε, και τα στοιχεία του ΩΣΑ και μερικές φορές ε, φαίνεται γνώμη την πραγματικότητα. Αυτό καλό θα ήταν να μελετήσουμε προσεκτικά τα στοιχεία. Και παρόλο που ελάχιστα ασχολούμαστε με το δημόσιο τομέα, οι κυβερνήσει Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσουν περισσότερα μέτρα για να, να προσλαμβάνουν και στο δημόσιο τομέα ε, μετανάστες και στις δυνάμεις ασφαλείας, ε, στις υπηρεσίες υγείας ή στη... στην εκπαίδευση. Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση και την κοινωνική επαφή. Επίσης, ε, θα δημιουργήσουμε πρότυπα σε διάφορους κλάδους και για τους μετανάστες, κάτι που συνέβη ήδη επιτυχώς σε μερικά κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, θα ήθελα να πω ότι ο οργανισμός μας έχει πραγματοποιήσει μελέτες σε περίπτωση ακραίας εκμετάλλευσης μεταναστών, εκεί που είναι οξύ το φαινόμενο της ακριβώς εκμετάλλευσης και θα μπορούσα να σας δώσω τελευταία στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα εθνικά προγράμματα σπουδών για να δούμε τι μαθαίνουν τα παιδιά για τους μετανάστες και πρόσφυγες, ιδιαίτερα στις χώρες που ε, δεν έχουν πολλούς πρόσφυγες ή μετανάστες. Ε, γιατί αναφέρεται η μεταναστες γιατι αναφερεται η συμμετοχη στην ιστορία των μεταναστών, σε χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης ε, ή στη Βουλγαρία, Ελλάδα και άλλες χώρες έχουμε μια πλούσια ιστορία μετανάστευσης και θα πρέπει να κάνουμε τον παραλληλισμό της αποδημίας τότε με τη σημερινή μετανάστευση. Επίσης να αποφύγουμε τις διακρίσεις ε, εις βάρος των μεταναστών και να εφοδιάσουμε τους δασκάλους καθηγητές να μπορούν να διαχειρίζονται διαπολιτιστικές συγκρούσεις και η καλύτερη ε, κατάρτιση και στις υποδομές και στο δυναμικό είναι η καλύτερη επένδυση για να αντιμετωπίσουμε την πολυμορφία ως ε, ατού και όχι ως πρόβλημα. Επίσης, ε, θα πρέπει όλα τα παιδιά να δημιουργούν δεξιότητες και γνώσεις με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και το καθεξής. Μόνο έτσι θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ε, συνύπαρξης με ε, μετανάστες από διαφορετική θρησκευτική η εθνοτική κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να μιμηθούμε τις καλές πρακτικές που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη και να τις γενικεύσουμε στα κράτη-μέλη και στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, ε, να λάβουμε υπόψη την διακήρυξη των Παρισίου του 2015 για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, στέγαση. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αποφύγουμε την ε, γετοποίηση στο στεγαστικό των ε, ε, μεταναστών, που είναι ένα φαινόμενο σε πολλές πόλεις, να καταρρύψουμε τους φραγμούς μεταξύ των κοινοτήτων, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση, με ε, κοινωνικές κατοικίες σε πολλές χώρες ε, και συμπερίληψη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό όπως έχει γίνει ε, σε πολλές πόλεις όπως στη Βιέννη. Μπορεί να αυξηθεί το πρόβλημα στο μέλλον γιατί πολλοί μπορεί να βρεθούν σε ένα νομικό κενό με τις σημαντικές ροές μεταναστευτικές το 2015 και 2016 και τέλος συμμετοχή και αρμονική συνύπαρξη. Πέρυσι το Δεκέμβριο, πριν από ένα μήνα δηλαδή, δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα σημαντική επισκόπηση για του μετανάστες και τι μειονότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντυπωσιακά αποτελέσματα και δείχνουν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών και των απογόνων του ε, νιώθουν με στενούς δεσμούς με την, χώρα στην οποία διαμένουν. 80% νιώθουν ότι ανήκουν στη χώρα αυτή και φαίνεται ότι εμπιστεύονται πολύ περισσότερο από το μέσο πληθυσμό ε, του δημόσιου φορεί. φορείς ε, ε, τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, για παράδειγμα. Επίσης, για, για τους μουσουλμάνους μετανάστες έχουμε έρευνα του Σεπτεμβρίου και σε αντίθεση με τα στερεότυπα, η έρευνα μας δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών και απαγόρων συμμερίζονται τις κοινές αξίες μας, ασθενίζονται τις κοινές αξίες μας, την ανεξιθρησκεία, το σεβασμό των διαφορετικών θρησκειών και εθνοτήτων, την ισότητα των φύλων, και ούτω καθεξής. Και μάλιστα η έρευνα μας δείχνει ότι εμπειρίες με ριζοσπαστικοποίηση και εξήμινηση χρέους έχει, έχουν μειωθεί στους δημόσιους, φορεί. στους δημόσιους φορείς. Και μάλιστα η δεύτερη γενιά μεταναστών έχουν πολύ ψηλά επίπεδα διάκρισης ε, και είναι θύματα ρατσιστικής βίας. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και να αντιμετωπίσουμε τη μυσαλλοδοξία και την ρητορική του μίσου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχής. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει πιο συστηματικά να εξορθολογήσουν πολιτικές για τους νέους μετανάστες και τους απογόνους των μεταναστών, για να αξιοποιήσουμε το, στο έπακρο το δυναμικό τους υπέρ των οικονομιών μας. Επίσης, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των μεταναστών στο δημόσιο βίο, ενεργό συμμετοχή στη συνδικάτα, για παράδειγμα, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ε, στις δημόσιες δουλεύσεις, αλλά και στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο. Φυσικά δεν υπάρχει μία θαυματουργή λύση για όλους, για όλες τις περιπτώσεις. Στην στο μεταναστευτικό και στο θέμα του ασύλου και της ένταξης. Ε, μπορεί να μην είναι ένα κουστούμι για όλους, αλλά μερικά κουστούμια είναι πολύ, καλύτερα ραμμένα από τα άλλα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα καλά κουστούμια, τις καλές πρακτικές, ε, να τις μιμηθούμε και να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση ως ευκαιρία και ως ατού και όχι ως πρόβλημα. Γιατί όπως δείχνει η επισκόπησή μας, ε, οι μετανάστες θα μείνουν εδώ σε εμά για πολλά χρόνια και καλό θα ήταν να του συντάξουμε όσο το δυνατόν συντομότερο, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση ουσιαστικά στα βασικά στοιχεία. Νομίζω ότι μας υπενθύμησε λίγο και τι νομοθεσία έχουμε και πόσο σημαντική είναι αυτή, αλλά δημιούργησε και το κατάλληλα κλίμα στο οποίο όλοι θεωρούν ότι μπορούν να συζητήσουμε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο ε, Κίμελ. Ε, ακούσαμε λίγα πράγματα για την εργασία ε, με τους Γερμανούς εργοδότες. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα έναν Γερμανό εργοδότη, ο οποίος θα μιλήσει για την εμπειρία του ως νέος Ευρωπαίος επιχειρηματίας, αλλά και άνθρωπος ο οποίος προσλαμβάνει νέους Ευρωπαίους και άλλους. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη... και ξέρετε, κυρίες και κύριοι, Πολλοί άνθρωποι τα τελευταία 100 χρόνια, πιο πολύ παραποτέ, για διάφορους λόγους έχουν προβεί σε μετανάστευση. Εγώ το 1973 έφυγα από το χωριό μου ε, στην ε, βορειοανατολική Τουρκία και πήγα στην ε, Κωνσταντινούπολη, στην Ισταμπούλ. Μετανάστευση δεν είναι κάτι το εύκολο. Το 1980 πήγα στην Γερμανία. Αυτή τη φορά γιατί η ενσωμάτωση ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Μάλλον αυτή τη φορά η ενσωμάτωση ήταν ακόμα πιο δύσκολη λόγω των γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών. Δύο φορές χρειάστηκε να ενταχθώ. Ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να βοηθώ τα άτομα που έχουν μεταναστεύσει για πολιτικούς ή οικονομικούς ε, λόγους. Ε, το 1993 ε, έφτιαξα την επιχειρήση μου, την Unipack, η οποία έχει ε, στο μεταξύ μεγαλώσει και έχει γίνει μια μικρομεσαία επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση. Πριν από 11 χρόνια δημιουργήσαμε το Hamburger Flaming, μια ένωση η οποία έχει ως σκοπό την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης. Όταν διαπιστώσαμε ότι Υπάρχουν και άλλες ενώσεις που ακολουθούν τους ίδιους ε, στόχους. Ε, δημιουργήσαμε τον, ε, την Ένωση BUV με το εξή λογότυπο. Ο BUV λοιπόν, η Ένωση αυτή, αυτή αυτός είναι ο ε, θέτει στο επίκεντρο την κοινοτομική ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών. Δίνει απαντήσεις στη δημογραφική αλλαγή, όπως είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με την ε, επίτευξη νέων αγορών. Κάποια παραδείγματα τώρα project και σχεδίων της BUV ε, παρουσιάζουμε στους μετανάστες στη Γερμανία. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε μαθητείες, προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις, για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Unity προέκυψε λοιπόν από την Ένωση του Κρατηδίου αυτού και έχει τους εξής ε, στην περιφέρεια, στις ε, ομόσπονδα κρατήδια ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνδράμει επιχειρήσεις και να αξιοποιεί τις εργασιακές δυνάμεις, ε, να αναπτύσσει διάφορα προγράμματα, να προαγάγει την ποικιλομορφία ως πλέον πλεονέκτημα της κοινωνίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας να ενισχύει με βιώσιμο τρόπο τις οικονομικές σχέσεις, γιατί θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί την καλύτερη ενσωμάτωση. Σε περίπτωση επιχειρηματικότητας ζουν ε, στο παλμό της καθημερινότητας ε, οι μετανάστες και παράγουν παραπάνω. Οι σημερινοί μετανάστες έχουν... είναι τυχεροί, γιατί τότε στην δική μου εποχή δεν υπήρχαν τέτοια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντική η στάση αντί των προσφύγων, γιατί θα πρέπει να μην υπάρχουν φόβοι, να γνωρίζουμε αλλήλους και μαζί να διαμορφώσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ουσιαστικά αυτό βοηθούμαστε όταν βοηθάμε τους ε, μετανάστες. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πιο πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς οι νέοι Ευρωπαίοι κατανοούμε πιο καλά τους ανθρώπους αυτούς, τους μετανάστες, από ότι οποιοδήποτε άλλη μέρη του πληθυσμού. Είτε μιλάμε για ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε για εθνικό επίπεδο. Αυτό που αποτελεί η καθημερινότητα είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Πριν από δύο χρόνια ε, προσέλαβα δύο Αφγανούς ε, μετανάστες με αντιεργασίας. Τότε λοιπόν κατάλαβα πολύ καλύτερα πως οι πρόσφυγες... Τι, τι αντίληψη υπάρχει για τους πρόσφυγες από τις εταιρείε, από τους εργοδότες, από το κράτος και τι, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Το πρώτο λοιπόν που κάναμε ήταν το εξή. Ένας συνάδελφος από την παραγωγή με τουρκικές ρίζες που ήταν υπεύθυνο για τους δύο αυτούς συναδέλφους, ε, μάλλον ήταν υπεύθυνο για όλα τα θέματα. Δεν μιλούσε παστού, αλλά προσπάθησε να, κάνει, να, να έχει μια επικοινωνία. Δεν είχε μόνο ευθύνη σε επαγγελματικό επίπεδο για του ανθρώπου αυτούς, αλλά και για καθημερινά ζητήματα, ιδιωτικά ε, ζητήματα. Ε, σε ποιο σχολείο να πάει το παιδί μου, πώς να μάθει η γενέκα μου γερμανικά, πώς θα πάω από το χ σημείο στο ψ σημείο. Οι επιχειρήσεις ε, που δηλώνουν ότι είναι διαθέσιμες να αφιερώσουν χρόνο και προσωπικό για την ένταξη των ε, προσφύγων, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από πόλεμα, από συγκρούσεις, προσπαθούν να φτιάξουν μια καινούργια ζωή εδώ, σε εμά. Το πρώτο που χρειάζονται είναι μια ανθρώπινη εγκύτητα, εμπιστοσύνη, φροντίδα, όχι γλωσσικά μαθήματα. Όχι πως δεν είναι σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της γλώσσας. Αυτό που θέλω να πω με πάσα σαφήνεια στην παρούσα φάση είναι ότι η εκμάθηση της γλώσσας δεν είναι δυνατό να προηγείται της ε, ανθρώπινης αντιμετώπισης. Γιατί συχνά γίνεται το λάθος στο εξή. Η επικοινωνία με τους μετανάστες αναβάλλεται. Περιμένουμε να μάθουν τη γλώσσα πρώτα. Νομίζω ότι η επιτυχία της Ένωσης Unity σε ό,τι αφορά την ε, απασχόληση των μεταναστών και των προσφύγων έγινε στο ότι ακούμε τους μετανάστες. Προσπαθούμε να τους καταλάβουμε ακόμα και αν δεν μιλάμε τη γλώσσα. Γιατί δεν ε, καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνουν πάντα οι άνθρωποι που μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά αυτοί που αισθάνονται τα ίδια συναισθήματα. και ρώτησα πριν έρθω εδώ να μιλήσω κάποιους ε, πρόσφυγες ε, αν θα ήθελαν να πούν κάτι στους πολιτικούς της Βρυξέλλες ε, και σας διαβιβάσω τα εξής μηνύματα. Τι είπαν. Είπαν λοιπόν, καταρχήν, καταρχάς, ανθρώπινη αντιμετώπιση ευγνωμοσύνη από καρδιάς. Όλα αυτά που μας έχουν λείψει στις πατρίδες μας, τις παίρνουμε εδώ από τους γείτονες, από τους συναδέλφους, από τον συνάνθρωπο. Αλλά αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε είναι τα παιδιά μας τα οποία μπορούν και πάλι να ζήσουν, να γελάσουν, να πάνε σχολείο. Είμαστε ευγνώμονες. Κατά δεύτερον, πολιτισμική κατανόηση. Εδώ η ενσωμάτωση δεν είναι δύσκολη γιατί ζούμε και κοντά με ανθρώπους από τους κύκλους μας. Ωστόσο είναι λιγότεροι αυτοί που ασχολούνται μαζί μας. Κατά τρίτον, το γλωσσικό εμπόδιο. Υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες που δίδονται για να μάθουμε τη γλώσσα θεωρητικά. Αυτό που λείπει όμως είναι οι πρακτικές ευκαιρίες και δυνατότητες κατά τέταρτον ε, με τα προσφυγικά, οι προσφυγικοί κατευλισμοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, οι ξενώνες συνήθω είναι καλοί, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει ο κόσμος στον ελεύθερο χρόνο του. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό γιατί μιλάμε για μήνες, χρόνια που πάνε χαμένα. Αυτή η απραξία μας καταστρέφει. Θέλουμε να είμαστε... Να, να δουλεύουμε, κάτι να κάνουμε, ακόμα και χωρίς αμοιβή, μέχρι ότου διευκρινιστεί το καθεστώς μας. Και τέλος, θα ήθελα να, να προσθέσω το εξής. Ε, θέλω να σας κάνω τις εξής προτάσεις. Καταρχάς, οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν πρόσφυγες και μετανάστες να τους προσφέρουν μαθητεία θα πρέπει να υποστηρίζονται πιο πολύ. Αυτή η υποστηρίξη μπορεί να είναι φορολογικά, πλεονεκτήματα, ε, προσωπικό παραπάνω, επιδοτήσεις, οτιδήποτε. Δεύτερον, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, εμπορικών επιμελητηρίων και ενώσεων εργαζοτών θα πρέπει να προσθεθεί πιο έντονα. Τρίτον, ΜΚΟ που δημιουργούνται από τους νέους Ευρωπαίους αυτούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν το σημείο επαφής μεταξύ επιχειρήσεων και προσφύγων. Ωστόσο, αυτές οι ΜΚΟ συνήθως δεν έχουν προσωπικό και δεν έχουν και πόρους. Μία από τις, ένα από τα καθήκοντα της Unity είναι να καταχωρήσει σε ένα κατάλογο αυτές τις ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να χορηγήσει πληροφορίες, γνώση και μακροπρόθεσμα να μπορέσει να τους καταρτήσει αυτές τις ΜΚΟ για να αποτελέσουν τη γέφυρα ακριβώς μεταξύ προσφύγων και επιχειρήσεων. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ και για τα όσα μας είπατε και για τα μηνύματα που μαζευάσατε και τις ε, συστάσεις ε, που είμαι βέβαιη ότι θα λάβει υπόψη το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε εθνικό επίπεδο λαμβάνουν καθήσεις αποφάσεις και όντως ε, η Unity είναι μια οργάνωση που είναι γνωστή και είχε επαφές μαζί μας στο Κοινοβούλιο και ήταν χρήσιμες αυτές τις επαφές. Θέλουμε προφανώς να συμπεριλάβουμε και εμπειρίες από το πολιτικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη. Εδώ έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση από την Πορτογαλία, από τη Σουζάνα Αμαδόρ. Ε, χρειάζομαι καλύτερα γυαλιά για να σας δω. Ε, έχετε 10 λεπτά. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα δηλαδή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την ε, διοργάνωση της πολύ σημαντικής αυτής διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για ένα πολύ επίκαιρο θέμα ε, και των Ηνωμένων Εθνών και των ε, κρατών μελών. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Πρόεδρο, τους καλεσμένους και κυρίως να ευχαριστήσω θερμά τον Οσμάν Κιμίλ που πραγματικά μας ενέπνευσε με την πολύ θετική του παρουσίαση για την ένταξη των ε, μεταναστών. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια άνευ κρίση και μεταναστευτικέ ροέ, χρειαζόμαστε ε, κοινή αναζήτηση ε, αϊφόρο λύσεων για τους μετανάστες και έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να τις βελτιώσουμε. Και απέναντι στην παγκόσμια δέσμευση για ε, να, βρούμε, να ξεπεράσουμε τα παλιά στερεότυπα και το φετελισμανισμό και να καταρρύψουμε τα εμπόδια που τους ε, τροφοδοτούν. Θα αναχαιτήσουμε τις κρίσεις αυτές και τα, τις ανθρώπινες τραγωδίες μόνο αν αποτρέψουμε ή προλάβουμε τις σειράξεις ε, και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο μέτρο που υπάρχουν τέτοιε κρίσει θα συνεχίσουν και αυτέ οι ε, αθρώε ε, ροέ των προσφύγων που χρήζουν διεθνού προστασία, γιατί οι χώρε του δεν μπορούν να εγγυηθούν την προστασία του ή είναι θύματα διώξεων. Επίση, από τη στιγμή που έχουμε υποδεχθεί ε, σε ασφαλεί χώρε στην Ευρώπη του πρόσφυγε αυτού, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την κοινωνική του ένταξη, που είναι και το σημερινό αντικείμενο τη συζήτηση. Γι' αυτό ε, χαίρομαι γιατί στι 20 Δεκεμβρίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κοινωνική και η κοινωνική και οικονομική εταίρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισαν την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Ένταξη, που θα δώσει νέε ευκαιρίε μετανάστε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενταχθούν στην αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έρχομαι στο παράδειγμα της Πορτογαλίας και την εμπειρία που είχαμε από την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Συνεχίζοντας το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, η κυβέρνηση ε, των σοσιαλιστών με υποστήριξη της αριστεράς υιοθέτησε μια ενεργό πολιτική ε, αλληλεγγύης για την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση στην Πορτογαλία προσφύγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 θεσπίσαμε μια ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο τη Μετανάστευση με πολιτικό συντονισμό από τον Υπουργό Εντουάρντο Καμπρίτα, ε, Υπουργό Εσωτερικής Διοίκησης. Έτσι έχουμε μια στρατηγική για την πλήρη ένταξη των ε, μεταναστών με βάση τις ακόλουθες αρχές ε, μια θεσμική, αποκεντρωμένη προσέγγιση με εταιρική σχέση, ολοκληρωμένη και αυτόνομη. Ε, και είναι ευθύνη του της ΥΠΑ ε, της Αρμοστίας ε, για, τις για τη μετανάστευση να βοηθήσει στην ενεργό ένταξη των προσφύγων. Θέλουμε επίση να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο στο θέμα των προσφύγων. Και γι' αυτό Έχουμε οργανώσει διάφορες εκστρατείες και στα σχολεία για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για την ανάγκη υποδοχής, φιλοξενίας και ένταξης των προσφύγων και μεταναστών. Επίση, έχουμε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με προτάσει για υποδοχή των προσφύγων και έχουμε εθνικέ ε, μονάδε στήριξη των μεταναστών και αρρωγή και ένταξη των μεταναστών, ενώ έχουμε και μία υπηρεσία τηλεφωνική μετάφραση, καθώ και το πρόγραμμα Πορτογαλικά για όλου. Έχουμε και επίση ένα πρόγραμμα e-learning μέσω του διαδικτύου για την εκμάθηση των Πορτογαλικών. Θέλουμε να στηρίξουμε την ένταξη των προσφύγων και τι ε, είναι σημαντικό γι' αυτό να συνεργαστούμε με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, και με τους θεσμούς υποδοχής. Και μάλιστα μετά την αρχική περίοδο 18 έως 24 μηνών μετά την ε, εισαγωγή έχουμε ενεργοποιήσει αυτού του μηχανισμού και έχουμε διάφορες, διάφορα επίπεδα. έχουμε μια ενημερωμένη παρακολούθηση των καταγραφών συνεργασία με τους φορείς που υποδέχονται τους ε, πρόσφυγες. Έχουμε συνοδεία κατά την άφηξη στο αεροδρόμιο, συνεργασία με τους φορείς υποδοχής. Στηρίζουμε τους φορείς ε, που διευκολύνουν την ένταξη και ούτω καθεξής. Στη διαδικασία αυτή έχουμε και την ε, συνοριοφυλακή και την υπετιαρμοστία που προσπαθεί να λάβει υπόψη τις ε, ανάγκες που ισχύουν και να, να κρατήσει αμύωτη την υποστήριξη προς τους φορείς υποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποδοχής και ε, ένταξης. Έχουμε και κατευθυντήριες γραμμές ώστε να λάβουμε υπόψη και την ατομική και την οικογενειακή ένταξη με λήψη υπόψη τους ε, εξής παράγοντες. Αποδοχή, εξέταση και μεταφορά των ετούντων, παροχή στέγης με θεσμική υποστήριξη, ατομική κατοικία, αξιοπρεπή, με, όλες, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καθημερινότητα, επίσης διατροφή, πρόσβαση στην υγεία, ψυχολογική υποστήριξη, πρόσβαση στην παιδεία, αναγνώριση των δεξιοτήτων, πρόσβαση στην πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ε, επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή στο κοινωνικό και δημόσιο βίο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ένταξη, νομική και δικαστική αρρωγή, κοινωνική βοήθεια, πρόθεση του διαπολιτιστικού και διαθρησκευτικού διαλόγου. Επίσης, για να εξασφαλίσουμε την αυτονόμηση ε, αυτών των ανθρώπων που υποδεχόμαστε στο, στην Πορτογαλική επικράτεια. Έχουμε μια ενεργό συμβολή των υπηρεσιών του θεματολογίου για την μετανάστευση μετά από τους 12 μήνες ε, άφεξης. Έχουμε επίσης ε, στην Λισαβόνα Πόρτο Κεφάρο δομές ε, στήριξης της ένταξης των μεταναστών και συνεργασία με το Ειδικό Γραφείο για την Αρρωγή και την Ένταξη των Προσφύγων. Και τηρούμε και τις αρχές που έχουμε αναλάβει, τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δείξει την, το ζήλο μας και την ε, προθυμία μας να υποδεχθούμε ε, πρόσφυγες με ανθρωπιστικές αξίες και με την ε, εγκάση υποστήριξη όλων των στρωμάτων της πορτογαλικής κοινωνίας. Και μάλιστα τα στοιχεία του 2017 δείχνουν ότι η Πορτογαλία στα πλαίσια της μετεγκατάστασης των εργαζομένων προώθησε την μετεγκατάσταση 1520 προσφύγων με τη συνεργασία πολυάριθμων δήμων με πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, την Ερυθρέα κυρίως. Επίσης, η συμμετοχή των δήμων ήταν ζωτική σημασία στη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, έχουμε συμμετοχή του επιμελητηρίου της Λισαβόνας, ε, Σύντρα, Πόρτο και ούτω καθεξής. Και μάλιστα είχαμε κατά 42% περισσότερες αιτήσει ε, φέτος από ό,τι πέρυσι. Και μάλιστα στην Πορτογαλία ε, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη γνώμη ότι θα πρέπει να βρούμε πολιτικούς και θεσμικούς ε, τρόπους που θα αποκλείουν τις πρωτοβουλίες κλεισίματος των συνόρων, θα διασφαλίζουν τη Συμφωνία του Σέγγεν και την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών των κρατών μελών. Θα προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα του χώρου ΣΕΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφοδιαστούμε με αποτελεσματικούς μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών κυρίως που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση από την κρίση. Στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο όλα τα κόμματα από, τα από τη αριστερά μέχρι τη δεξιά τάχθηκαν υπέρ της πράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της ε, πιστής εφαρμογής αρχής ε, της Συνθήκης Γενέβης του 1951, του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί αυτό είναι το καθήκον μας ως ανθρώπων και ως ε, πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, σημαντικοί δείκτες ε, του προγράμματος αυτού. Θα πρέπει να ληφθούν ως δείκτες η υγεία, η γλώσσα, η παιδεία, η νομοποίηση, αριθμός γεννήσεων, αριθμός ένταξης, ε, ενημέρωση και απασχόληση. Με βάση την έκθεση αξιολόγησης πολιτικής υποδοχής της Πορτογαλίας του Δεκεμβρίου του 2017, ο τομέας της υγείας έχουμε μεγάλη ένταξη 100%, 98% στην παιδεία και ε, οι πρόσφυγες, τα παιδιά των προσφύγων έχουν πρόσβαση 100% σε όλα τα σχολεία της Πορτογαλίας. Μερικές φορές ε, απλώς οι οικογένειες προτιμούν να κρατήσουν τα παιδιά μέχρι τα 5-6 χρόνια. Ε, επίσης ε, έχουμε 560 πολίτες σε ενεργοδράση που έχουν ήδη βρει απασχόληση. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενή τομέα έχουμε 25% και 50% στο τριτογενή τομέα. Στον δευτερογενή τομέα γύρω στο 25%. Θέλουμε επίσης ε, τις δράσεις ε, στήριξης των τεχνικών υποδοχής και ένα σχέδιο που έχει στόχο την ε, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των προσφύγων, την δημιουργία ε, ε, επαγγελματικών ευκαιριών σε συνεργασία με τους εργοδότες και με τις πορτογαλικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουμε μόνο θετικά στοιχεία, δεν έχουμε μόνο τέλεια ένταξη. Υπάρχουν και περιορισμοί που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά αυτού του περιορισμού θα του καταπολεμήσουμε. Πάντω, τα συνολικά αποτελέσματα του προγράμματο είναι αρκετά θετικά και είμαστε υπερήφανοι γιατί βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Και όπω είπε ο Αντώνιο Κουτιέρε, κάθε φορά που υποδεχόμαστε πρόσφυγε, ουσιαστικά συναντούμε την ανθρωπιά μα και ε, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ ε, πλήρης εικόνα του τι ακριβώς κάνετε και είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα έρχουν ερωτήσεις και ε, θα μιλήσουν και μαζί σας και μετά το πέρας της εκδήλωσης γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο κράτους μέλους, ε, στη ρίζα δηλαδή. Και για να προσθέσουμε και δύο λόγια ακόμα, να περάσουμε στον τελευταίο μιλητή μας ε, σε αυτό το πάνελ. Έχουμε τον εισηγητή από την Επιτροπή των Περιφερειών για πέντε λεπτά, τον κύριο Καλογερόπουλο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πάρω αφορμή από την κυρία από την Πορτογαλία. Είδαμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα σε μια χώρα όπου ο Πρωθυπουργό της, ο Κώστα, ήταν δήμαρχος Λισαβόνας και σαν αυτοδιοίκηση είχε προωθήσει αυτές τις δομές. Σας λέει σήμερα λοιπόν η κυρία από την Πορτογαλία ότι και η δεξιά και οι σοσιαλιστές και η αριστερά δεν μαλώνουν για το θέμα αυτό, αλλά έχουν σύμπνια. Εν αντιθέσει με άλλα κράτη που είναι η προμετωπίδα για να κερδίσουν τις εκλογές. Πέταξε μακριά τους μετανάστες για να γλιτώσει η χώρα μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ουσία. Χαίρομαι πάρα πολύ κυρία μου διότι πραγματικά και η εξαποστάσεως εκμάθηση της γλώσσας της Πορτογαλικής για να σέβονται οι μετανάστες τους κανόνες, να γνωρίζουν τους νόμους, να διαβάζουν τους νόμους της Πορτογαλίας και να εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά και η εκπαίδευση της γλώσσας. Πώς είναι δυνατόν να μιλήσεις ή να ενταχθείς σε ένα κοινωνικό σύνολο όταν δεν μιλάς τη γλώσσα ακόμα και των γονιών προκειμένου τα παιδιά όταν γυρίζουν από το σχολείο να έχουν συνεννόηση στην καινούρια πατρίδα που βρίσκονται. Χαίρομαι επίση που ο κύριο, ο φίλο μα εδώ, ο γείτονα από την Τουρκία, ο κύριο Κιμίλ, καταξιώθηκε στη Γερμανία. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί από μόνο του κατάφερε να επιβιώσει όπω πολλοί μετανάστε από την Ελλάδα ή από την. πηγαίνανε στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Σήμερα δυστυχώ φεύγουν λόγω τη οικονομική κρίση και τη δυσκολία που υπάρχουν και πολλά φωτεινά μυαλά πάνε πάλι στην Ευρώπη και δουλεύουν γιατί έχουν καλύτερου μισθού η μετανάστευση θα υπάρχει πάντα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μην χάσουμε το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, ανθρώπων και ιδεών και τον πολιτισμό της. Η συνθήκη της Σέγγεν δεν πρέπει να ακουμπηθεί. Εκείνο που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή σαν Επιτροπή Περιφερειών, γνωμοδοτικό όργανο μετά τη Λισαβόνα, είναι ο ρόλος τοπικών αρχών στην ενσωμάτωση των προσφύγων. Γι' αυτό προηγουμένω στην κυρία Κουτήρα που ήταν εδώ μιλήσαμε για του πρόσφυγε. Απλά. Θέλω να σα πω το εξή. Ω πού θα πάει αυτή η εμπορία των ανθρώπων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και βεβαίω σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν κάποιοι κανόνε. Και αυτό πάει να κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών, να πει την άποψή τη, δηλαδή οι τοπικέ οι, τοπικές, οι δήμοι και οι περιφέρειε, τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι όμω είναι υπόθεση των, των Εθνικών Κοινοβουλίων εάν θέλουμε να είμαστε μια Ευρώπη ενιαία, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου, να μπει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Αν ο καθένας κάνει κατά το δοκούν, λέγοντας άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε, τότε αυτό δεν λέει τίποτα. Να μην επανέλθω ότι όπως είναι οι Ουκρανοί που πάνε σήμερα στην Πολωνία, εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνοί ερχόντουσαν στην Ελλάδα, είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν χριστιανοί, για να το επιβεβαιώσουμε δεν ήταν μουσουλμάνοι, κύριε Χίνγκη, ή ακόμα και Ρώσοι που ερχόντουσαν ή απόγονοι Ελλήνων από τη Ρωσία, αυτοί ενσωματώνονται, ε, ενσωματώνονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε πολέμους, η κλιματική ρωσια αυτοι ενσωματωνονται μεσα σε μικρο χρονικο διαστημα τωρα κατά τον κύριο Τραμπ που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σε λίγο διάστημα η Μεσόγειος θα έχει γίνει Αφρική και η Αφρική δεν θα υποφέρεται. Θα έχουμε άλλα κύματα μετανάστευσης, αλλά πάμε στα σημερινά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν τι λέμε. Ότι οι πύλες εισόδου εκείνες που υπάρχουν θέλουν βοήθεια. Και θα πρέπει να καταλάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται το θέμα, ότι εκείνοι οι οποίοι υποδέχονται τους μετανάστες, μιλάνε με τα επιμελητήρια, δεν πρέπει να, υπά... πρέπει να βρίσκουμε δηλαδή τόσο ένα, έναν κύριο κοιμήλ για να μπορεί να, να πάρει τους μετανάστες στην εργασία. Αν αυτοί δεν ενσωματωθούν και έχουν μόνο τη βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται μαρτζινέ. Δεν μπαίνουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι απέναντι. Και δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια εκείνους οι οποίοι είναι για το, για το άσυλο μετανάστες και εκείνοι οι οποίοι είναι οι λαθρέοι οικονομικοί μετανάστες. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Και τι ζητάμε. Ζητάμε στελέχη, τεχνικά στελέχη που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πύλες εισόδου για το άσυλο για να μην αμφισβητείτε ποιο είναι, ε, είναι ή όχι διότι σήμερα υπάρχει αμφισβήτηση. Εγώ πέρασα από Γερμανία και μου εξετάσαν το διαβατήριο, επειδή έρχονται πολλοί μετανάστες στην Ελλάδα, αν είναι αυθεντικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αν αυτή η Ευρώπη με τη μορφή την ανοιχτή της Σέγγεν ισχύει για όλους. Και το λέω αυτό γιατί και η Γερμανία βρέθηκε στη Δίνη και άλλα, και άλλα ευρωπαϊκά κράτη με το θέμα το μεταναστευτικό. Πόσοι λαϊκιστέ ή οι εξτρεμιστές δεν το χρησιμοποιήσαν σαν ασπίδα για να κερδίσουν την ψήφο των συμπολιτών τους. Ο φόβος και ο τρόμος. Ποιοι? Τα ανθρωπάκια που τα πνίγουμε στη Μεσόγειο. Έρχεται λοιπόν η αυτοδιοίκηση σήμερα και λέει τα παιδιά πρέπει να μάθουν γράμματα των μεταναστών, άρα πρέπει να μάθουν τη γλώσσα. Και ο ίδιο και οι μετανάστε. Εάν έχουν δεξιότητε, πρέπει να τι χρησιμοποιήσουμε και να του εντάξει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, η Δήμη στην κοινωνία εργασία και να βρουν κάποια δουλειά ώστε να είναι χρήσιμοι. Να συνεισφέρουν από τα, τις, τις, τα, τα ταμεία τα οποία θα πληρώνουν κιόλα για την υγεία η οποία θα του παρέχεται να είναι ενεργοί πολίτε για να μπορούν να ενσωματωθούν. Και το λέω αυτό όχι μόνο για του Δήμου τη Μεσογείου, το λέω και για του Δήμου των άλλων κρατών, των βορείων κρατών. Διότι οι δήμαρχοι που δεν είναι εκεί, εμεί συμφωνούμε, σα πληροφορώ, στην εισήγηση που κάνω, έχω μόνο τέσσερι τροπολογίε. Του πιέζουν πολλέ φορέ οι μόνιμε αντιπροσωπείε του δημάρχου να ακολουθήσουν την τακτική τη εθνική κυβέρνηση. Δηλαδή μακριά. Ο δήμαρχο όμω, επειδή είναι ένα από εμά, είναι η Ευρώπη, ο άνθρωπος, η κοινωνία των πολιτών των Ευρωπαίων σου λέει ρε φίλε για κάθισε. Εμείς αυτοί είναι συνάνθρωποι μας. Αφού μπορώ να του βρω μια δουλειά εγώ, δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Εκεί όμως πρέπει να κοιτάξουμε ορισμένες ιδιαιτερότητε που υπάρχουν. Δηλαδή το γλωσσικό, αυτό που είπατε το πολιτιστικό, το πολιτισμικό, γιατί σας έχετε άλλο, άλλη διαδικασία. Το θρησκευτικό, εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία. Και έρχεται σήμερα λοιπόν οι φίλοι μας από την Πορτογαλία και μας λέει μια δομή που υπάρχει. Εγώ δεν θυμούμαι όταν ήμουν δήμαρχος το 2007 ότι είχαμε φτιάξει κέντρο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και εξ για τους μετανάστες για να μπορούν να ενταχθούν. Γιατί τότε η εισήγησή μου ήταν για την ένταξη, τις καλές εντάξεις. Ο δε πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας ήταν υπουργό εσωτερικών, ο Παυλόπουλος, τότε. Ο οποίος έφτιαξε το πρώτο κέντρο που υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα στη Μυτιλίνη, στο Μορέα Δυναμικό των 3.000 ανθρώπων και είναι 10.000. Σε λίγο θα είναι περισσότερο από του κατοίκου. Αυτό λοιπόν ενώ πέρσι τρει γυναίκε από τη Μυτιλίνη ήταν να πάρουν το βραβείο Νόμπελ, μεγάλε γυναίκε, γιατί βοηθούσαν του μετανάστε, σήμερα ακούμε τα εξαμάξει ότι υπάρχουν ιδιότητε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αποσυμφορηθεί. Εδώ έρχεται λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφέρειες να δώσουν το χέρι βοηθεία. Εάν οι εθνικέ κυβερνήσει θέλουν να παίρνουν τα χρήματα και να τα παίζουν κατά το δοκούν είναι πρόβλημα και δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα. Επίσης οι ΜΚΟ, οι οποίες είναι εξαιρετικές, πρέπει όμως να ελέγχονται για τα χρήματα που παίρνουν και την αποδοτικότητα που έχουν στις ενέργειες που έχουν κάνει. Ποιος τις ελέγχει, κανένας. Τι επικοινωνία έχουν με τους δημάρχους και τις τοπικές αρχές, καμία. Δηλαδή μιλάνε με την Ευρώπη και δεν μιλάνε με τους ντόπιου. Αυτά λοιπόν είναι οι παράμετροι τις οποίες βάζουμε. Και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με καλύτερο τρόπο. Εγώ άκουσα και βουλευτές από την Πολωνία και τους σέβομαι. Διότι φανταστείτε ότι από τα πρώην κομμουνιστικά κρατία, από την, την περιοχή της Ουκρανίας που γίνεται ο, ο μεγάλος χαμός, πόσες χιλιάδες άνθρωποι πάνε. Ναι, είναι ένα, μετα, ένα μεταναστευτικό κύμα. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά πρέπει να δούμε, να βάλουμε κανόνες. Και πρέπει να βάλουμε κανόνες γιατί εμείς είμαστε πολίτες, δεν νομοθετούμε, Ακολουθούμε τη διαδικασία, είμαστε σύνομοι, αλλά έχουμε και φωνή. Τι λένε αυτοί οι κανόνε, Ή όλοι ακολουθούμε τη διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενοι βέβαια τα εθνικά μα δίκαια και τα συνταγματικά, αλλά όχι όπου μα βολεύει. Και όπου δεν μα βολεύει φεύγουμε. Διότι εδώ στον ανθρώπινο πόνο και στο θάνατο και στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε λιμπεράλε. Υπάρχει ο άνθρωπος αυτό λέει η αυτοδιοίκηση. Κλείνοντας αγαπητοί φίλοι, για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, θέλω να σας πω ότι αυτό το σχέδιο που χρειάζεται πρέπει να ακολουθεί από όλους. Εάν δεν το ακολουθήσουμε, τότε με συγχωρείτε, εγώ δεν δέχτηκα ποτέ να πάω υποψήφιο βουλευτή γιατί μου έκανε η αυτοδιοίκηση. Ήμουν δήμαρχο, ήμουν νομάρχη. Δεν θέλω να πάω βουλευτή, βράδελφέ μου. Με ικανοποιεί η Επιτροπή των Περιφερειών. Θέλω όμω να σα πω, επειδή σα σεβόμαστε και επειδή νομοθετείτε, σκεφτείτε την Ευρώπη και όχι την επόμενη εκλογή σα. Σα ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά θα ε, καταλάβουν καλά. Περνάμε τώρα στις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έχουμε περίπου 20 λεπτά γι' αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε συγκεκριμένοι. Πολύ θα το εκτιμήσω. Και ξεκινάμε με μία ακόμα ελληνική παρέμβαση. Thank you, Madam President. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη κτίστηκε πάνω σε ένα πλαίσιο συνενέσεων, συμβιβασμών και υπερβάσεων από τα κράτη-μέλη, προκειμένου πλέον πρόσβαση στην πληροφορία η γεωγραφική θέση επηρεάζει καθοριστικά. Η απόσταση μερικές φορές οδηγεί σε αποστασία. Αυτό κάναμε στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στοιχείο καλής ναυτοσύνης, είναι και το στοιχειοδός ανθρώπινο καθήκον μας. Από εκεί και πέρα βέβαια προκύπτουν υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι η επιτάξη διαδικασιών χορήγησης ασύλου ώστε να υπάρξει γρήγορη διάκριση μεταξύ προσφύγων που μάλλον θα μείνουν και παρατύπων μεταναστών που θα επαναπροωθεί στην αγορά εργασίας προσφύγων μεταναστών. Τρίτον, και τελειώνω, υλοποίηση σχεδίου απασχόληση με ευθύνη και προτάσει κράτου μέλου σχετικά με ευκαιρίε τη χώρα μου, τη επιφύλαξε τη μοίρα να σηκώσει δυσανάλογα μεγάλο βάρο του προβλήματο. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, σαφώ μπορούμε και καλύτερα. Ένα πλέον τελικά στον κοινό τόπο. Σα ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και ζητώ συγγνώμη που έκανα λάθος το όνομα. Ε, κοίταζα το πρόγραμμα. Περνάμε σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, στην Νορβηγία. Η Κριστίν Γιάνσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να παρέμβω. Κάποιες παρεμβάσεις από την Νορβηγία που είναι συνδεδεμένο κράτος και μέλος της Σέγγεν. Εμείς ε, παρακολουθούμε τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ε, στενά και λάβαμε πάνω από 30.000 γραμμα και έχουμε υποδεχθεί μετανάστες από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρατηρήσεις μου όμως ε, για την ένταξη ε, είναι ότι είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία και απαιτεί δέσμευση και από τις δύο πλευρές, ε, όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από η ανεργία στην πρώτη γενιά των μεταναστών είναι τριπλάσια του ευρύτερου πληθυσμού στην Νορβηγία. Και όσον αφορά τα παιδιά της πρώτης γενιάς των μεταναστών, ε, υπάρχει πρόβλημα, κυρίως μεταξύ των γυναικών και πολλά παιδιά εγκαταλεί προγράμματα ε, ε, για ε, εξέβριση θέσης εργασίας και εκμάθηση γλωσσών είναι δύο χρόνια, αλλά ε, Τέσσερι στους δέκα μόνο ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο και βρίσκουν μια θέση εργασίας. Η απασχόληση λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας και ε, θέλουμε τα αυτά. Συμφωνώ ότι η ένταξη θα πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε ε, μετανάστη. Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο το πλαίσιο και να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν και ε, πρότυπα για τις γυναίκες και νομίζω κάτι που δεν ακούστηκε σήμερα, προγράμματα κοινωνικών επιδεμάτων θα πρέπει να συνδέονται πιο στενά με τη δυνατότητα εργασία του καθενό. Το μήνυμά μα πρέπει να είναι απόλυτα σαφή. Το κράτο πρόνοια δεν είναι βιώσιμο εάν οι μετανάστε ε, δεν έχουν θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ ιδέες, όπως είπατε και εσείς, ε, για τη δική σας τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ε, καλό θα ήταν να είμαστε σε επαφή ε, με όλα όσα ακούμε σήμερα, για να δούμε κατά πόσον υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, ε, ιδιαίτερα κατά τον επόμενο ευρωπαϊκό ε, προγραμματισμό, την επόμενη προγραμματική περίοδο. Να περάσουμε τώρα στους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό. Σε σχέση με αυτά που είπε η συμπατριώτησα μου Σουζάνα Μαντόρ για το ρόλο της Πορτογαλίας και τη σημασία που έχει της ε, διαδικασίας ένταξης, υποδοχής πρώτα και ένταξης των προσφύγων. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω και αναφυσβήτητα υπάρχουν εξαιρετικά ικανοποιητικοί δείκτες για την υγεία, για την πρόσβαση στην παιδεία, για τη φίτηση των παιδιών, για την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Στην ε, Πορτογαλία τα πανεπιστήμια είναι αυτόνομα και υπάρχουν πολλές πτυχές της ευαισθητοποίησης, ε, της διαδικασίας της μετεγκατάστασης που αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτία τη άρνησης μερικών χωρών μελών να συμμετέχουν στην γενική αυτή αλληλεγγύη και να δεχτούν δίχτυα των λαθροδιακινητών που χρησιμοποίησαν μερικές φορές στη διαδικασία της μετεκατάστασης ε, για να βρουν πύλη εισόδου από άλλες χώρες. Φυσική μετανάστευση, το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, γι' αυτό ακριβώ και θα πρέπει να την χάνει κατάλληλη ρύθμιση και πρέπει να είναι ισορροπημένη και να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των χωρών, τα συμφέροντα των ε, ανθρώπων. Φυσικά. Κύριε Χέλγα ναι, δεν είναι εδώ στην παρούσα φάση, ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε απαντήσεις από το πάνελ, γιατί είμαι βέβαιο ότι θα υπάρχουν και θέματα τα οποία χρήσουν διευκρίνησης. Ο κύριος Λίμπεκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω κάποια σημεία, αν μου επιτρέπετε. Καταρχά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε από διάφορε γωνιέ του ακροτηρίου η σημασία τη κατηγοριοποίηση και τη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών. Αυτό νομίζω μα βρίσκει όλου σύμφωνου. Έστω και αν υπάρχει ένα πράγμα επί το οποίο συμφωνούμε. Ένα από τα μεγάλα λάθη που κάναμε ήταν να αποκαλούσουμε όλους που κατέφτασαν πρόσφυγες. Και ξέρουμε ότι ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων δεν έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε και τους όρους που χρησιμοποιούμε. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο αυτό το παράδειγμα της Αυστραλίας, του Καναδά και είναι μέρη του ΩΣΑ, άρα έχω αρμοδιότητα να μιλήσω και για αυτού λίγο. Ε, οι χώρες αυτές προφανώς έχουν πολύ έντονη διαχειριζόμενη μετανάστευση και ανάλογα προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πάντα επιτρέπουν ε, σε όλη την οικογένεια να καταφτάσει. Αυτό είναι το μήμα του πακέτου, μιας και μίλησαμε προηγουμένως ε, την οικογενειακή επανένωση. Είναι λοιπόν πολύ ανοιχτή αυτή η πολιτική τους. Έχουν επίσης προγράμματα επανεγκατάστασης έχουν αντίληψη του ότι άμα ότι προσελκύουν του, το, το, τους πιο υψηλά εκπαιδευμένους, αλλά έχουν αυτή τη λογική της επανεγκατάστασης. Προτείνουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη να τα υποστηρίξουμε στην όλη διαδικασία ένταξη, γιατί νομίζω ότι όταν επενδύουμε χρήματα στη γλωσσική εκπαίδευση, για παράδειγμα, υπάρχουν αποτελέσματα. Ένα πράγμα, για παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους μετανάστες. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αποτέλεσμα ήταν να φτάνει κανείς στο επίπεδο Β1 στο ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο για την εκμάθηση των γλωσσών. Όταν φτάνει λοιπόν κανείς στο Β1 είναι πολύ μεγάλο το αντίκρισμα. Μετά από εκεί και πέρα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι φαίνεται. Και τέλος, να κλείσω με ένα μια φλόγα ελπίδα, γιατί μαθαίνουμε για τις διαφορές και έτσι στην εργασία μας ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιαζόμαστε σε δείκτες για τη διαφορά μεταξύ των μεταναστών και των ε, αυτοχθόνων. Αυτό που μας ε, προκαλεί μεγαλύτερο, μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι σε πιο πολλές περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ των διαφορών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγαλύτερη από την διαφορά μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων στην κάθε χώρα. Ένα στοιχείο επίση, ε, το οποίο φαντάζομαι θα μας έβρισκε όλους σύμφωνους και το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε για να προσδοκούμε τις μετανάστες είναι να ακολουθούν του κανόνες της εκάστοτε χώρας. Και ξέρουμε από τις έρευνες ότι είναι και το μόνο το οποίο πραγματικά... Στη Γερμανία, ο και Κιμίλε, έχουμε στη Γερμανία το μισθό. Για όλου. Μετανάστε, πρόσφυγε αλλά και για τους ε, ντόπιου, τους Γερμανούς. Υπάρχει δηλαδή ε, ο μισθός ανά ώρα, ο οποίος καθορίζεται από την αγορά και ισχύει για όλους. Άρα, αυτοί οι κανόνες στηρούνται. Δεν μπορεί κανείς να απλά να τους αγνοήσει. Από αυτή την οπτική και προς την κατεύθυνση αυτή μίλησα όταν είπα ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό που με απασχολεί εμένα βασικά είναι να έχουν θέσεις μαθητείας, πρακτικής. Προκειμένου να τους χορηγούνται δεξιότητες και γνώση και βάσει της γνώσης αυτής και της δεξιότητας αυτής να βρουν μια θέση εργασίας στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το καθοριστικό και για μας. Θα ήθελα λοιπόν αυτή η βάση να μπορούσε να ίσχυε για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παύλου. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα σχόλια στη συζήτηση και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων και στοιχείων. Όπως είπε και ο Τόμας, όλες οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες ε, ε, οπιτών ε, δεν αντανακλά την πραγματική τους γνώμη και την επιθυμία τους να εντάξουν τους μετανάστες σε κοινέ αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε τελική ανάλυση η κοινωνική ένταξη είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα θεμελιωδών αρχών και συμφώνησαν να αναπτύξουν πολιτικές όχι μόνο επειδή, όχι επειδή είναι υποχρεωμένα γιατί είναι... Πολίτες ποιος θα διώξει τους πρόσφυγες. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ο άνθρωπος. Και πιστεύω ότι πέρα και πάνω από όλε τι διαδικασίες εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν γιατί έχουν μια χρονική διάρκεια που λειτουργούν χωρίς να κάνουν ενδιάμεσες εκλογές που μπορεί να πάει ο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να ασχοληθεί, να ενταχθεί, να νιώσει ότι είναι χρήσιμος εκεί που πήγε, να κάνει εκμάθηση της γλώσσας, να τον βοηθήσουν, είναι οι δήμαρχοι και οι περιφέρειες. Εξάλλου αυτή είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη των Δήμων και των Περιφερειών. Η Ευρώπη αυτό ό,τι θέλετε. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Με την έννοια, όχι την εθνική μας πατρίδα. Θέλετε να την κρατήσουμε ορθιά. Γιατί είναι προσχηματικό αυτό τώρα από τους πρόσφυγες. Θα έχουμε άλλα θέματα. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη έδινε όπλα στη σύραξη που γινότανε. Κρατήσουν τον πληθυσμό τους στη Βόρεια Αφρική. Τώρα λοιπόν λέμε να το κάνουμε. Εμείς οι φουκαράδες που ήταν αυτοδιοικητικοί το λέγαμε μια δεκαετία πριν. Βοηθήστε τους για να μην λακίσουν όπως λέμε στην Ελλάδα. Να μην τρέξουνε. Εκεί η ανθρώπινη ύπαρξη δεν μετράει τίποτα. Αντί μα που φεύγουν ήδη έτοιμα και αποδυναμώσουν, θα βγουν νέα παιδιά. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Ξαναγυρίζει στον τόπο από όπου προέρχεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Να βοηθήσουν δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν την άμεση... Πολύ εύκολο, προσέξτε με, είναι πολύ εύκολο να πας σε μια χώρα όπου έχει δυσκολίες με το μεταναστευτικό και να πολιτευτείς εις βάρος του μεταναστευτικού. Το είδαμε σε διπλανά κράτη. Πώς ακραίες οργανώσεις μπήκανε σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν κάθομαι να κάνω αυτή την κριτική. Ούτε τις προσωπικότητες. Είδαμε και τον Brexit στην Αγγλία τι έγινε. Τα παιχνίδια λοιπόν μπορεί να υπάρχουν τα πολιτικά και τα για τους στρατηγικά, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Ελληνός τροπαέζε, καραμίκο. Ελληνός τροπαέζε. Σας ευχαριστώ από τη ρίζα άνθρωπους που δουλεύουν με τους πολίτες και όλοι εμείς να συνεργαζόμαστε. Δεν θα σχολιάσω τα νόητα παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί ραγίζει η καρδιά μου της Επιτροπής ε, Λίπετη την Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, για αυτό το τελευταίο πάνελ, την καταληκτική συζήτηση, χρειάστηκε να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, ε, γιατί τελικά ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ήρθε στο πρώτο τμήμα της συζήτησης και θα δεν θα μπορέσει να είναι εδώ για την ε, καταληκτική συζήτηση. Έχουμε όμως εδώ τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον κύριο Αμπρόζη μαζί μας, ο οποίος εκπροσωπεί το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε τις συζητήσεις που κάναμε σε ένα πιο παγκόσμιο πλαίσιο, στην προετοιμασία του Παγκόσμιου ε, Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Μετά από την ε, παρέμβασή σας θα ξεκινήσει η συζήτηση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Νομίζω Είχατε μια πολύ γεμάτη ημέρα. Συζητάμε την ε, νόμιμου διάβλου μετανάστευση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει και να προσδώσω ένα πλαίσιο στο διεθνές επίπεδο, όπως ακούστηκε, ε, εντός του οποίου γίνεται η εφαρμογή του εθιματολογίου και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ε, λίγο καλύτερα τι προϋποθέτει αυτό για την εφαρμογή του. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη από το 2015, δηλαδή από τότε που είχαμε το θεματολόγιο, το διεθνές ε, ε, σενάριο έχει αλλάξει και έχει αλλάξει ε, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Καταρχάς, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, η μετανάστευση έχει πρωταρχικό ρόλο για την ε, ανάπτυξη της ε, μετανάστευσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2016 ενέκρινε και την ε, δήλωση της Νέας Υόρκης η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία ε, της ανάπτυξης δύο παγκοσμίων συμφώνων έναν ε, ε, για τη μετανάστευση και στη δήλωση της Νέας Υόρκης ε, είχαμε τις βασικές αρχές και τα βασικά πρότυπα τα οποία συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν σημασία όχι μόνο γιατί έχουμε δύο καλά έγγραφα που περιλαμβάνουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά και ε, γιατί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και η δήλωση της Νέας Υόρκης περιλαμβάνουν δεσμεύσεις από πλευράς ε, διεθνούς κοινότητας, περιλαμβάνουν πρότυπα και αρχές που κάθε χώρα που έχει προσπογράψει αυτά τα δύο έγγραφα και όλες ε, οι χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν προσπογράψει, ε, δεσμεύονται να τηρήσουν και να σεβαστούν αυτές τις ε, δεσμεύσεις. Για μας εδώ στην Ευρώπη και για όλους εσάς που προσωπείτε και χώρες που έχουν υπογράψει αυτές τις δεσμεύσεις, σημαίνει ότι όταν συζητάμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη μετανάστευση, τις νόμιμους διάβλους, την ένταξη και τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά, μας δεσμεύουν οι ε, υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει στο διεθνέ επίπεδο στην ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μα δεσμεύουν όχι μόνο γιατί έχουμε προσπογράψει αυτέ τι δεσμεύσει, αλλά και γιατί ε, αν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να συνεχίσουν να είναι ισχυρό παράγον στο διεθνέ προσκήνιο θα πρέπει να τηρήσουν τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει, να είναι αξιόπιστοι και να τηρήσουν αυτέ τι δεσμεύσει με αξιοπιστία και να διατηρήσουν και την εμπιστοσύνη ενώπιον των υπολείπων μελών της διεθνούς κοινότητας. Ότι αυτό που έχει συμφωνηθεί δηλαδή θα μεταφράζεται και ε, σε απτά αποτελέσματα τι σημαίνει αυτό για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, τους νόμιμους διάβλους ε, ε, και την νόμιμη μετανάστευση. Και τα δύο έγγραφα και οι δύο διαδικασίες που σας ανέφερα και οι βιώσιμοι στόχοι και το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, αναφέρονται στην βελτίωση των νομίμων διάβλων μετανάστευσης ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μετανάστευση και η μετανάστευση μπορούν να είναι κάτι χρήσιμο για την ανάπτυξη και την οικονομική αναβάθμιση και των κοινοτήτων καταγωγής και των κοινοτήτων προορισμού και φυσικά και για τους ίδιους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε κατά την εφαρμογή του θεματολογίου μέχρι τώρα, ένα θεματολόγιο το οποίο ε, είναι ένα αρκετά ισορροπημένο έγγραφο, ευθύ εξ αρχή περιλαμβάνει τέσσερι πυλώνε, οι οποίοι αναφέρονται ε, στα θέματα τη βελτίωση των νομιμών διάβλων και την καταπολέμηση τη παράτυπη μετανάστευση, ε, την πρόθεση και την αναβάθμιση των κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τμήμα της στρατηγικής ε, του θεματολογίου και αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει μια υπερβολική εστίαση σε ένα συγκεκριμένο πυλώνα, ο οποίος έχει σχέση με την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των επιστροφών, αλλά δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στους άλλους πυλώνες και πιο συγκεκριμένα στον πυλώνα που αφορά την ενίσχυση των νομίμων διάβλων. Και η συζήτηση που γίνεται από τότε που δημοσιεύθηκε το θεματολόγιο για τη μετανάστευση και ε, κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί, τι σημαίνει νόμιμη διάβλος, ε, ε, νόμιμος διάβλος για αυτόν που φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε Αυτό είναι κάτι σημαντικό το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα ισορροπία στην εφαρμογή ε, του θεματολογίου για τη μετανάστευση, λαμβάνοντας υπαλλήσουμε ότι ε, ξέρουμε σαφώς ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρώπη και αυτέ οι διάφορε κατηγορίε ε, προποθέτουν όταν θα χρειάζεται και να φροντίσουμε ότι θα γίνει η ένταξη. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα αυτό είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε σοβαρά μηχανισμούς, πολιτικές και προγράμματα, τα οποία θα οδηγήσουν και σε διαρθρωτικές αλλαγές ε, ε, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό ο κινητήριος μοχλός είτε δικαιολογημένα είτε ίσως και υπερβολικά ήταν ε, ε, η απάντηση στην κρίση. Σε κάποιο βαθμό μας φόβησε ο αριθμός των αφήξεων και η αντίδραση ε, ήταν ε, αυτή που θεωρούσαμε κατάλληλη για απάντηση σε μια κατεπίγουσα κατάσταση. Αλλά πλέον δεν είναι κατεπίγουσα κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι ε, ότι φτάνει ένα πολύ μικρό κλάσμα των μεταναστών ε, που κινούνται ανά τον κόσμο. Δεν είναι κρίση, δεν είναι κατεπίγουσα κατάσταση λόγω συγκεκριμένων συνδικών. Είναι ένα διαρθρωτικό ζήτημα. Και είναι ένα διαρθρωτικό ζήτημα που υπαγορεύεται από κάποιες ε, πολύ ε, σαφές, σαφείς διαστάσεις που βλέπουμε και στην Ευρώπη αλλά και στη γειτονική περιοχή, ιδιαίτερα στην Αφρική. Η πρώτη σαφής απόδειξη της διαφορετικής κατάστασης είναι η δρομογραφική κατάσταση στην Ευρώπη ε, που ε, έχει συνεχή μείωση ε, και δεν το λέω εγώ, το λέει η Eurostat, Ευρωπαϊκό όργανο που λέει ότι η δημογραφική καμπύλη στην ε, Ευρώπη μειώνεται με κάποιες εξαιρέσεις σε κάποιες χώρες, αλλά σε γενικές γραμμές μέχρι το 2050 οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε Μείωση της τάξης του 18% της δημογραφικής καμπύλης. Ε, ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε αντίθετες τάσεις. Επομένως ε, αυτές οι δύο συνιστάμενες ε, δυνάμεις ε, θα πρέπει ε, ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε αντίθετες τάσεις. Επομένως αυτές οι δύο συνιστάμενες δυνάμεις θα πρέπει Για να το πω με απλά λόγια, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε αρκετούς εργαζομένους για να καλύψουν το κενό της αγοράς εργασίας που θα διαθέτουν τα συστήματα με νόμιμο, ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει πολιτική κλειστών θυρών. Εάν κλείσουμε την πόρτα δεν μπαίνει κανείς και οπότε είμαστε ασφαλείς. Πρώτον, δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ρίως, μια υπερβολικά κλειστή πολιτική ε, και η παντελής απουσία αυτή τη στιγμή σχεδόν ε, θα ήταν στο σύστημα VIS, ε, το σύστημα θεωρήσεων, θα ήταν ταυτοποιημένη. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους και δεν μπορούμε να την γνωρίζουμε γιατί δεν υπάρχει καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε καθώς ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα το οποίο διαθέτουμε. Να ακούσω σχόλια και ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Αμπρόζη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους εθνικούς βουλευτές ότι αν θέλουν το λόγο θα πρέπει να κάνουν ένα νεύμα. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Outside, then... Ναι. Μάλλον βγήκε έξω. Άλλος κανείς. Outside, then... Ναι. Μάλλον βγήκε έξω. Άλλος κανείς. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Κανείς. δεν για πρώτη φορά το λόγο, αλλά πραγματικά θα ήθελα να πάει χαμένη ευκαιρία και σε αυτή την τελική φάση της νέας αυτής ε, διακοινοβουλευτικής διάσκεψης που τηρεί τις ε, διατάξεις της Λισαβόνας, καλό θα είναι να εκμεταλλευτούμε κάθε λεπτό και στην προηγούμενη την εναρμόνιση και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των λύσεων. Αυτή είναι η μόνη λύση. Εναλλακτική δεν υπάρχει. Και επίση θα πρέπει να αλλάξουμε την εστίασή μας φαινόμενο της σφαιρικής αντίληψης και κατανόησης της μετανάστευσης. Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει την αποτυχία, τη μέχρι τώρα αποτυχία της ευρωπαϊκής της ε, εξώθησής της πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των συνόρων της ε, και με τίμημα ε, κάποια την ασφάλεια. Κακός. Γιατί μερικές φορές η μετανάστευση γίνεται ο δούριος ύπος του, της τζιχαντιστικής από ανθρώπους που ήταν γέννημα θρέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπης. Και όσοι κάνουν το αμάλγαμα μετανάστευση και τραυματίζεις των μεταναστευτικών ρόν. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το εργασιακό δυναμικό της ε, ε, συνεισφοράς ε, στις κοινωνικές υπηρεσίες, χάρη στην δική μας συνεισφορά και την συνεισφορά των εθνικών βουλευτών. Αυτά, γιατί βρισκόμαστε με κάποια συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Τάνια Φαγιό, νομίμων διάβλων πρόσβαση των μεταναστών. Κύριε Αμπρόζη, μήπως θα θέλατε να σχολιάσετε αυτά τα ενδιαφέροντα σχόλια των συναδέλφων. Λίγα σχόλια για αυτά που ακούσαμε και